Να ξαναρχίσουμε αν θέλετε καθίστε. So you can hear. Θα το γυρίσω στα Ιταλικά, οπότε αν θέλετε φορέστε τα ακουστικά σας. Ευθύς αμέσως να καλωσορίσω τους προστακλημένους μας, τους εμπειρογνώμονές μας που έχουν ήδη καταφτάσει Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που η Επιτροπή μας σήμερα έχει διοργανώσει αυτή τη σημαντικότατη ακρόαση για ένα θέμα που για μας είναι κεντρική σημασία και γίνεται όλο και πιο κέρια σημασία για την υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή την ένταξη των προσφύγων και των παιδιών τους μέσω της κατάρτισης και της παιδείας. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά γενικότερα για παιδεία και πολιτισμό. Δύο μορφές πλήρους ένταξης Ξέρουμε ότι υπάρχουν ανεπίσημες και επίσημες αρμοδιότητες σήμερα, αλλά αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε τα θεμέλια μιας συμμετοχικής και πολυφωνικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που μπορεί να δώσει σάρκα και οστά σε μια πραγματική ιδιότητα του πολίτη με συμμετοχή στα πολιτιστικά, στην κοινωνική ζωή πριν από τις νομικές ε, Έχουμε μια δραματική ανθρωπιστική κρίση σήμερα σε εξέλιξη. Δυστυχώς πλήττει και την Ευρώπη, ε, όχι μόνο εκτός των σύνορων της Ευρώπης, αλλά και εντός. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν τραγικές μορφές περιθωριοποίησης και πολλές φορές μη εξωπρεπείς συνθήκες υποδοχής παιδιών, γυναικών και προσφύγων. Νομίζω ότι ως Κοινοβούλιο σωστά έχουμε καταβάλει εντατικές προσπάθειες για να εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την μετανάστευση και να διαρθρωθούν περισσότερο ε, σωστά τα πρότυπα ε, υποδοχής και ένταξης των προσφύγων και θυμίζω ότι ακόμη και έναντι της παρουσίας ε, μιας ανίποτης μαζικής προσέλευσης προσφύγων με ανηλίκους και γυναίκες να είναι το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ αυτών ε, θυμίζουμε ε, με επιμονή ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα προηγούνται τη ηθαγένεια και ότι ακόμη και αν δεν αναγνωριστεί το καθεστώ του πρόσφυγα, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, στην μέρημνα την αξιοπρεπή διαβίωση και την προστασία των ανηλίκων. Εδώ πρέπει να γίνονται σεβαστέ και διεθνεί συμβάσει και για το άσυλο και για του ανηλίκου και την προστασία του και για τα ανθρώπινα δικαιώματα που δυστυχώ σήμερα δεν μου φαίνεται ότι στην Ευρώπη το πραγματοποιούμε. Είναι, είμαι λοιπόν ιδιαίτερα ευτυχή που σήμερα βρίσκομαι εδώ δίπλα σε μία συνάδελφο, την Κασετού Κιέντζε, η οποία είναι η εισηγήτρια μια σημαντικότητα της έκθεσης στην Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη και επίσης πληρωτήρα μέλος στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων γιατί θέλουμε να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση στις πολιτικές ένταξεις των προσφύγων, ιδίως ε, σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο. Ε, ε, ήταν σημαντικό να το διευκρινίσω αυτό γιατί την απόφαση για αυτή την ακρόαση τη λάβαμε μαζί με τους ε, συντονιστές των διαφορών πολιτικών ομάδων ώστε καθώς θεωρήσαμε αναγκαίο, ε, ενώ η Επιτροπή για τις Ελευθερίες του Πολίτη συζητά το θέμα αυτό, η Επιτροπή η Επιτροπή συζητά ε, η Επιτροπή Έμπλη μάλλον με την κυρία Μπονιφέη Συγήτρια συζητά το θέμα της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας και υπάρχει και η δική μου έκθεση. Θέλουμε να καλύψουμε λοιπόν περισσότερε από μία προσεγγίσει. Η μία είναι αυτή που θα λέγαμε τη ανάδυση, του κατεπήγοντο μάλλον. Του κατεπήγοντο και τη μεγάλη πίεση που δέχεται η Ευρώπη και το τι θέλουμε να διασφαλίσουμε ω προ την πρόσβαση στα εκπαιδευτικά ε, ιδρύματα σε αυτή τη φάση, την κατεπίγουσα, απασχοληθήκαμε εδώ στο Κοινοβούλιο και ζητήσαμε να διπλασιαστούν οι πόροι για να προσφερθούν εκπαιδευτικέ υπηρεσίες στους ανηλίκους. Όχι μόνον ε, έπειτα, ε, αλλά και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εδώ και στους καταβλισμούς των προσφύγων και υπό τις συνθήκες αυτές της κατεπίγουσας. Και έπειτα καθίσταται σαφές ότι τα άτομα, ξένοι, αλλοδαποί μετανάστες, θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο πλήμα της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οπότε αυτή τη στιγμή αντιπαραβάλλονται περισσότερο από ό,τι ποτέ τα διάφορα μοντέλα, οι διαφορετικές εμπειρίες που έχουν ε, συλλέξει οι εμπειρογνώμονές μας με τους οποίους θα συζητήσουμε, μοντέλα ένταξης, συμμετοχής, αξιοποίησης της παρουσίας αυτών των αλλοδαπών και ελπίζω και δυνατότητας να καταλάβουμε ότι πρόκειται για πλούτο, ανθρώπινο πλούτο, μια νέα ανθρώπινη ομάδα για την Ευρώπη. Για αυτό το σκοπό λοιπόν σήμερα έχουμε αυτήν την ομάδα προσκεκλημένων κοντά μας. Θα σας δώσω με τη σειρά το λόγο. Ε, ε, ξεβονίμων έχω την ε, κυρία Κιέντζε, τον κύριο Πιατσεντίνη από τον ΟΑΣΕ, ο οποίος παρακολουθεί τις εκθέσεις του, του για τα θέματα της εκπαίδευσης και σε αυτό θα επικεντρωθεί και στην ε, ομιλία του. Ιδίως ό,τι αφορά την γλωσσική ένταξη, την εκμάθηση γλωσσών, Επίσης τη δόκτορα Μπριζίτε Μπάλμπακ, η οποία είναι ε, σχολική διευθύντρια στην ε, νότια Ρινανία Βεσφαλία και είναι μέλος και της ομάδας των ε, δασκάλων. Έπειτα έχουμε την κυρία Έμπελ, Μελανή Έμπελ από το ε, Συμβούλιο Νέων του Βραδεμβούργου, την κυρία Έλενα Μπεζότσι, Ιταλίδα εκπρόσωπο της Επιστημονικής Επιτροπής του, Ιδρύματος, ε, του Διεθνούς Ιδρύματος για τους, για τους μετανάστες και μετά την κυρία Μαριάν Πονσλέ και την, την κυρία Πατρίς Βίχερς από, την, ε, από το Διεθνές Ίδρυμα για τη Χουντή Μενουχήν. Ε, και η ίδια είναι μετανάστηδα η οποία έχει εγκατασταθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Θα, δώσουμε, λοιπόν, θα ακούσουμε και τη δική της φωνή για το θέμα αυτό. Έχουμε επίσης πολλές ομάδες Έχουμε, με συγχωρείτε, έχουμε και άλλους προσκεκλημένους, αλλά δεν βλέπω ποιοι είναι. Α, είναι τέσσερις. Τέσσερις μόρ, Ο κύριος Μόργανο από την Ιταλία έχει προσκαλέσει μια ομάδα επισκεπτών και έχουμε και... Με συγχωρείτε τώρα τα ονόματα στα χέρια μου και 7 προσκεκλημένους της ε, κυρίας Κέντ οι οποίοι προφανώς βρίσκονται εδώ γιατί ενδιαφέρονται για την όλη συζήτηση. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Να δώσω το λόγο στη Σασίλ Κέντ. Σα ευχαριστώ που βρίσκεστε εδώ και θα δώσω το λόγο και στην κυρία Κινίτση από την Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη για το θέμα τη διαδικασία. Ευχαριστώ τη για την σοβαρή τη δουλειά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Σίλβια. Με... Είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σήμερα εδώ για να ε, παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης πρωτοβουλίας για τη Μεσόγειο και την σφαιρική μας προσέγγιση, την ε, προσέγγιση στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Ε, ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να παρουσιάσω εδώ τις σκέψεις μου και να συζητήσω για αυτές μαζί σας. Όπως γνωρίζετε, βρισκόμαστε στην παραμονή της ψηφοφορίας, διότι εμείς θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή Ελευθερίων του Πολίτη αύριο το πρωί και η Επιτροπή θα τοποθετηθεί ακριβώς για το κείμενο αυτό, που επιτρέψτε μου να το πω, ε, μεταφράζει σειρά μηνών δουλειά και επίσης την ε, δυνατότητα συμφωνίας μεταξύ πολλών πολιτικών ομάδων. Όχι απλώς καταλήξαμε λοιπόν σε συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων, αλλά υπήρξε ε, ο καρπός συλλογικής δουλειάς. Ξεκινήσαμε από ένα σαφές γεγονός αναντήρητο. Το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι τόσο περίπλοκο που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να το διαχειριζόμαστε με μέσα και πολιτικές διαδικασίες που χρησιμοποιούσαμε ως σήμερα. Οι πολιτικέ που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία 20 χρόνια και σε επίπεδο ένωση και σε επίπεδο κρατών μελών έχουν ξεπεραστεί. Χρειάζεται λοιπόν μια προσέγγιση της ασφάλειας στα πλαίσια αυτής της κατεπίγουσας ε, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και εν ώψη των λαμβάνοντα μάλλον υπόψη τις αλλαγέ που υπάρχουν εδώ μεταξύ καμία πολιτική ως τώρα δεν φάνηκε ικανή να εμποδίσει την μετακίνηση πληθυσμών από τη Μεσόγειο ή τα Βαλκάνια, ότι θα συμβεί αυτό στο μέλλον. Έτσι λοιπόν πρέπει η τα βαλκανια ούτε θα συμβει αυτο στο μελλον ετσι λοιπον πρεπει η ευρωπη να το δει αυτό μια ευκαιρία για την μελλοντική της ζωή. Υπάρχει μεγάλη μετακίνηση πληθυσμών, είναι μεγαλύτερη μετακίνηση ανδρών και γυναικών μετά τη Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πρέπει να εξετάσουμε το μεταναστευτικό αυτό φαινόμενο και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι ακριβώς και το νόημα του σχεδίου έκθεσης που συνέταξα για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη να υπάρξει μια σφαιρική προσέγγιση. Ήθελα να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε με αυτήν την ιδιαιτερότητα, αλλά σιγά σιγά όλη η κατάσταση ε, κατέληξε να είναι κατεπίγουσα. Χρειάστηκε λοιπόν να ε, συμπεριλάβουμε και την οδό των Βαλκανίων όπως έλεγα, οι προσπάθειες διατησίας διαμεσολάβησης για να γεφυρώσουμε τις διαφορετικές απόψεις μας οδήγησε σε ένα κοινό κείμενο με συγκεκριμένε συστάσεις σε διαφορετικούς τομείς όπου θα μπορούσαμε να παρέμβουμε. Το κύριο μήνυμα που εκφράζει η έκθεση είναι ότι το φαινόμενο τη μετανάστευση δεν μπορεί να αναχαιτιστεί, αλλά πρέπει να γίνει αντικείμενο διαχείριση μέσω όλων των πολιτικών μα και των πολιτικών μέσων που διαθέτουμε. Αυτό πρέπει να γίνει με την βέλτιστη δυνατή ε, με τον ευθυγράμμιση τη εξωτερική πολιτική με την πολιτική ασφάλεια και τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, θεσμικών και μη. Το σχέδιο έκθεση προτείνει συγκεκριμένε δράσει, βραχυπρόθεσμε, μεσοπρόθεσμε και μακροπρόθεσμε. Και διαρθρωτικές πολιτικές ε, που σκοπό έχουν να ε, καλύψουν το φαινόμενο αντιμετωπίζοντας τα γενεσιουργά του αίτια, δηλαδή τις ρίζες του προβλήματος, τους λόγους για τους οποίους ε, οι μετανάστες γίνονται μετανάστες, μετακινούνται. Η έκφραση αλληλεγγύη σημαίνει πλήρη κατανομή των ευθυνών. Αυτά όλα δεν μπορούν να παραμένουν θεωρητικέ ε, σκέψει και έννοιε, αλλά πρέπει να λάβουν σαρκά και σωστά ε, στο σχεδιασμό τη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική. Ξεκινώντα λοιπόν από αυτά τα δύο ε, σημεία που εκφράζονται και στο άρθρο 80 τη Συνθήκη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να προχωρήσουμε υπάρχει και η απαραίτητη νομική βάση για την μελλοντική υλοποίηση και πρόβλεψη νομοθεσίας. Η αλληλεγγύη πρέπει να εκδηλωθεί για τις κατεπήγουσες καταστάσεις που ζούμε σήμερα μέσω της πλήρους στήριξης σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης. Ε, ταυτόχρονα ζητάμε από τα κρατημέλη να ε, προβλέψουν έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό ε, διαρκή που να ασχολείται, να αφοσιωθεί μάλλον ε, στην έρευνα, τη διάσωση και την αντιμετώπιση συνθήκων κινδύνου και να χρηματοδοτείται επαρκώ και από την άποψη τη πρικοδότησή του τη δημοσιονομική αλλά και των μέσων που θα διαθέτει. Η αλληλεγγύη όμω δεν είναι μόνο η διάσωση στη θάλασσα. Η αλληλεγγύη εκφράζεται και με την προσφορά ελπίδα σε όσου προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο, το λοιμό και τι διώξει. Πρέπει λοιπόν να του δώσουμε και μια εναλλακτική στη ζωή τους εφόσον ε, ξεκινάνε αυτόν τον ε, διάπλου. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε το μηχανισμό επανεγκατάστασης, να γίνει ένας υποχρεωτικός ε, μηχανισμός για τους ετούντες άσυλο εντός της Ένωσης. Ένας μηχανισμός που στο βαθμό του δυνατού θα λαμβάνει υπόψη και τις προτιμήσεις των ετούντων ανάλογα με τη χώρα προορισμού τους. Όμως εκφραστήκαμε και υπέρ ενός μηχανισμού δεσμευτικού, μόνιμου, για την ε, ε μετεγκατάσταση ενός μεγάλου αριθμού του των ασύλου ε, εντός των κατωμέλων. χωρίς να παραμελήσουμε ε, άλλες εκφράσεις αλληλεγγύης, όπως οι ανθρωπιστικές μας ε, δράσεις ή οι θεωρήσεις οι ανθρωπιστικές το να διαχειριστούμε συνετά το φαινόμενο της μετανάστευσης σημαίνει ότι θα ανοίξουμε διάβλους, νόμιμες οδούς μετανάστευσης, γιατί η Ευρώπη θα μπορέσει να ε, προχωρήσει μόνο να αξιοποιήσει τα προσόντα των ανθρώπων αυτών που καταφτάνουν η έλλειψη εργατικού δυναμικού ε, μέχρι τώρα με ψηλά επαγγελματικά προσόντα είναι μια σημαντική, ένα σημαντικό στοιχείο. Πρέπει να αναθεωρήσουμε όλες τις πολιτικές μετανάστευσης και τις, να δούμε και τις οικονομικές μας ανάγκες. Πρέπει να δούμε ακριβώς την είσοδο και την εγκατάσταση εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες με νέο τρόπο. Σε ό,τι αφορά την οικονομική μετανάστευση καταδικάζουμε ε, με πυγμή ε, κάθε ε, εργασιακή εκμετάλλευση των ε, νεοαφιχθέντων, διότι εφόσον τα κάτι μέλη έχουν λάβει τέτοια μέτρα, Ουσιαστικά αυτό ισοδυναμεί με εμπορία ή δουλεμπόριο. Είναι απαραίτητη η πλήρη η πληρης εφαρμογη τη Οδηγία 52 του 2009 που προβλέπει την προστασία των θυμάτων εμπορία ή διακίνηση ανθρώπων με ερευνητικέ δραστηριότητες και δικαστικέ διαδικασίες. Χρειάζεται επίσης αναθεώρηση της γαλάζιας κάρτας, της Blue Card, μια φιλόδοξη βέβαια πρόβλεψη, που όμως χρειάζεται για την ένταξη στην αγορά εργασίας όλων των καθών μελών. Όμως, εφόσον ανοίξουμε διάβλους, οδούς νόμιμες για την άφηξη των μεταναστών στο ευρωπαϊκό έδαφος, θα πρέπει έπειτα να υπάρξει και η θέσπιση μέτρων, μέτρων φιλόδοξων, με φιλόδοξες πολιτικές, που σκοπό θα έχουν πρώτα απ' όλα την ένταξη ένταξη που αφορά ε, όλος ιδιαίτερος και την Επιτροπή σας. Η ένταξη των μεταναστών κατά πρώτον και κατά δεύτερον η ελεύθερη κυκλοφορία των προσφύγων. Νομίζω ότι η ένταξη είναι το σημείο κλειδί ακριβώς για την επιτυχία όλων των πολιτικών μας. Για μια μελλοντική πολιτική μετανάστευση που θα είναι κοινή. Η πρόκληση που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να καταρτήσουμε μια προσέγγιση που να ε, ασχολείται κατά προτεραιότητα με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ένταξή του στον κοινωνικό ιστό, τον οικονομικό ιστό, αλλά και τον πολιτιστικό ιστό τη χώρα που του υποδέχεται. Πρέπει να εξασφαλίζονται δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα να προβλέπονται και υποχρεώσει, ε, παρόμοια με αυτά των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν ω προ την ένταξη το σχέδιο έκθεσης ε, έχει εκφραστεί λιγότερο αλλά συμπεριλάβαμε και αυτή τη διάσταση χάρη στι τροπολογίε που υποβλήθηκαν και που προήλθαν και από τη δική σα επιτροπή από τους βουλευτές της Επιτροπής Πολιτιστικών Υποθέσεων. Καταφέραμε λοιπόν να ενισχύσουμε τη διάσταση αυτή που εκπροσωπεί αναπόσπαστο, θεμελιώδες τμήμα της μεταναστευτικής πολιτικής που θα είναι κοινή. Τι συμβαστικέ τροπολογίες έχουμε κυρίως ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να προβλέψουν πολιτικές ένταξης για τους πολίτες των τρίτων χωρών, μέτρα που θα πρέπει κατά κύριο λόγο να ασχολούνται με την ε, ένταξη και όχι την, τον αποκλεισμό. Επίσης υπογραμμίσαμε το γεγονός ότι είναι σημαντικός ο ρόλος που θα ε, αναλάβουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, διότι η ένταξη αρχίζει ακριβώς από, την, ε, το τοπικό επίπεδο. Πρέπει να προβλεφθούν συγκεκριμένα προγράμματα ένταξης Ζητήσαμε από τα κάτι μέλη να ε, περάσουν στους ε, πρόσφυγες δυνατότητα να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους στη χώρα υποδοχής τους και θα πρέπει να προβλεφθεί γι' αυτό η διάθεση στέγης, πρόσβαση στην εκπαίδευση, η δυνατότητα να ε, παρακολουθήσουν μαθήματα επαγγελματική κατάρτιση και γλώσσα και βεβαίω να ενθαρρυνθεί ο διαπολιτιστικό διάλογο. Να σημειώσουμε εδώ το βασικό εργαλείο ένταξη είναι η εργασία. Ακούσαμε ότι υπάρχει έκθεση πρωτοβουλίας και για την εργασιακή ένταξη των ε, μεταναστών και γι' αυτό, εντάξει, ε, και γι αυτό καλέσαμε και τα κρατημέλη να εφαρμόσουν σωστά το άρθρο 15 της οδηγίας υποδοχή των μεταναστών που προβλέπει την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Δεν θα ήθελα να ε, παρατείνω την αναμονή σας, διότι το αποτέλεσμα που εκφράζεται με το σχέδιο έκθεσης είναι, ε, μια, ε, είναι καρπός ενός έτους εργασία, εργασίας. Αύριο θα ψηφιστεί λοιπόν Και ελπίζουμε ότι θα είναι θετικό το αποτέλεσμα και η έκβαση, διότι είναι τόσο περίπλοκο το φαινόμενο αυτό που μόνο εφόσον συνδυάσουμε διάφορε πολιτικέ κινήσει και κατάλληλα εργαλεία θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν να ξεφύγουμε από τη λογική του φόβου. Το Κοινοβούλιο δείχνει ότι αναλαμβάνει τις ευθύνες του ε, έναντι του φαινομένου αυτού και των αιτιών που τον προκαλούν. Ζητώ λοιπόν να προσπαθήσουμε να παροτρύνουμε τα κρατημέλη για να εγκαταλείψουν τις εγωιστικές τους τοποθετήσεις ε, και το κλείσιμο των συνόρων ενώ πρέπει να αφοσιωθούν στο να θέσουν τα θεμέλια μιας πραγματικής κοινή μεταναστευτικής πολιτικής. Βλέπω ότι έχετε στα χέρια σας το σχέδιο έκθεσης. Δεν ανέπτυξε όλα τα σημεία γιατί ξέρω ότι υπάρχουν κάποια τμήματα που ενδιαφέρουν όλες ιδιαίτερα στην Επιτροπή σας. Ευχαριστούμε Σεσίλ για την ε, κατανόηση, αλλά έχουμε πίεση χρόνου και κυρίως αύριο θα είναι σημαντική μέρα γιατί έτσι καλλιώς η ψηφοφορία στη Λίμπε είναι αύριο. Βλέπουμε ότι έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά. Είδαμε τι προσοχή σε άκουσαν όλοι και πόσο συμμεριζόμαστε την ανάγκη των ε, μεταναστών ε, να ε, ληφθούν σοβαρά υπόψη οι ανάγκες τους. Πρέπει να πω ότι είναι πολλοί συνάδελφοι τη Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και εγώ η ίδια, που αποστήλαμε τροπολογίε στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και ευχαριστώ γιατί πολλέ έγιναν δεκτέ παράδεκτες μέλλον και κυρίως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, τα εκπαιδευτικά πρότυπα, η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση και ακόμα και αυτό το σημείο του ψηφίσματος που είχε περάσει για τους ε, πρόσφυγες τον Νοέμβριο. Δηλαδή εκπαιδευτική διάδρομη που οδηγούν στα ανώτατα ιδρύματα για τους ε, πρόσφυγες από εμπόλεμη κατάσταση χώρες που γίνονται δεκτοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το μεγάλο θέμα που θα μπορούσαμε από τη μια να την ονομάσουμε κατεπίγουσα κρίση και από την άλλη ε, αυτό το κύμα αφήξεων που δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση προσωρινό Όλα αυτά θα πρέπει να καταγραφούν μεταξύ των πώληση των πολιτικών που προσπαθούν να υλοποιήσουν διάφορα κατημέλια αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε τι συστάσεις μπορούν να εκφράσουν σχετικά η Επιτροπή αλλά και το Κοινοβούλιο για το γενικό θέμα της ένταξης των προσφύγων, των νέων και των ανηλίκων μέσω του πολιτισμού. Ας τώρα στην ουσία της συζήτησή μας να δώσω αυτή αμέσω το λόγο στον ε, δόκτορα Πιατσαντίνη του ΟΑΣΕ που θα μας παρουσιάσει τις δικές, του, τις δικές της σκέψεις. Good, afternoon everyone. I'm Mario Piacentini. I'm a... Καλό σας απόγευμα. Είμαι ο Μάριο Πιατσεντίνη αρμόδιος του προγράμματος του ΩΣΑ για τις ε, ε, προοπτικές αυτές και ευχαριστώ για την πρόσκληση να σας προσφωνήσουμε για αυτό το σημαντικό θέμα. Στην δική μου παρέμβαση θα σας δείξω κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν τι γίνεται σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία όσον αφορά την ένταξη των νέων προσφύγων. Το κύριο σημείο μου είναι ότι το σχολικό σύστημα αντιδρώντας σε αυτά τα θέματα πρέπει να έχει τεράστια εμβέλεια κοινωνικά άσχετα από την, ε, το σκηνικό προσφύγων. Ο πληθυσμός των προσφύγων έχει αυξηθεί εντωμεταξύ από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης και είναι και πιο πολυσχηδής. Και σύμφωνα με τα στοιχεία μας το 2012 12% είχαμε ε, από αυτό το ποσοστό και είχαν γεννηθεί στο, στην Αλοδαπή. Μεταξύ 2003-2012 το ποσοστό των προσφύγων μαθητών στα σχολεία μας αυξήθηκε από 4 6% σε ποσοστίες μονάδες. Σε κάποιες χώρες όπως την Ισπανία, Ιταλία, Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, και διακυμάνσεις στις ίδιες τις χώρες οι πρόσφυγες μαθητές ε, συνήθως βρίσκονται στις ίδιες τάξεις και στα ίδια σχολεία και αυτό αυξάνει την, πρόκληση να ενταχθούν ε, αυτά τα παιδιά στο σχολικό σύστημα και από πλευράς του εκπαιδευτικού προσωπικού. Δημοσιεύσαμε αυτή την έκθεση που είναι ε, το τίτλος είναι <clears throat> «Παιδιά προσφύγων στα σχολεία μας, αντιμετώπιση της πρόκλησης που ε, έχουμε ενώπιόν μας» και αυτή η έκθεση έχει συλλέξει στοιχεία από βάσει δεδομένων για την ανάλυση των ε, επιδόσεων των παιδιών προσφύγων στα σχολεία τους. Τα στοιχεία δείχνουν με σαφήνεια ότι η εκπαίδευση και ο πολιτισμός των παιδιών προτού ε, γίνουν μετανάστες ε, έχει σαφή επίπτωση στις επιδόσεις τους. Όμως οι επιδόσεις τους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών υποδοχής. Συγκρίνουμε <clears throat> σε σχέση με τις επιδόσεις τους ε, των μαθητών που γεννήθηκαν σε αραβόφωνες χώρες και τις συγκρίνουμε τις επιδόσεις με άλλους μαθητές. Στην Ολλανδία έχουμε καλύτερες επιδόσεις από ό,τι στη Δανία, στην Φινλανδία ή στο Κατάρ. Βλέπουμε δηλαδή τις διαφορές σε σχέση με τα παιδιά από αραβόφωνες χώρες που βρίσκονται στην Ολλανδία και είχαν υψηλότερους βαθμούς στα μαθηματικά από τους άλλους και αυτό όχι μόνο εξαρτάται από τις επιδόσεις τους αλλά εξετάζουμε επίσης και το κοινωνικό περίγυρο και την κοινωνική ένταξη των παιδιών στα σχολεία. Ένας δείκτης ε, της ικανότητας να εντάξουν τα παιδιά στις κοινωνίες ε, είναι το να έχουν το αίσθημα ότι ανήκουν σε αυτά τα σχολεία, σε αυτό το, στον περίγυρο τα παιδιά. Σε αυτό το γράφημα έχουμε το ίδιο ουσιαστικά το οποίο προηγούμενα είδαμε συγκρίνοντας το αίσθημα του πώς ανήκουν τα παιδιά από αραβόφανες χώρες ε, αν αισθάνονται ότι ανήκουν στον σχολικό περίγυρο και στις κοινωνίες τους. Έχουν καλύτερες επιδόσεις ως προς αυτό στην Φινλανδία υψηλότερος βαθμός ε, ε, αίσθησης του ότι ανήκαν σε αυτόν τον περίγυρο σε σχέση με την σύγκριση για παράδειγμα των άλλων που βρισκόντουσαν σε άλλες χώρες. Τα στοιχεία μας επιβεβαιώνουν ότι η ψυχολογική ευημερία και των, παιδιών αυτών δεν ε, προέρχεται μόνο από τον πολιτισμό στις χώρες τους, ε, χώρες ε, προέλευσης, αλλά διαμορφώνεται και από τα σχολεία και τις κοινωνίες μας όταν βρίσκονται αντιμέτωπα αυτά τα παιδιά με την ε, διαδικασία μάθησης ε, και, την, και βιώνουν ε, τον περίγυρό τους. Στο επόμενο γράφημα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε ένα από τα θέματα που αναλύουμε στην έκθεση και είναι ένα από τα κύρια στοιχεία των, της κοινωνικής και σχολικής ένταξης των παιδιών στις κοινωνίες μας. Και είναι ο συντελεστής της γλώσσας, ο παράγοντας της γλώσσας που μαθαίνουν και χρησιμοποιούν στα σχολεία τους. Ξέρουμε ότι πολλά παιδιά προσφύγων αντιμετωπίζουν αυτόν τον φραγμό, το πρόσκομα της γλώσσας. 64, 64 ε, από 64% ε, των μαθητών αυτών μιλούν μια διαφορετική γλώσσα από ε, εκείνη που είναι η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν και βλέπουμε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούν μια, το, μεγαλύτερο, κατά το μεγαλύτερο διάστημα μια άλλη γλώσσα. Οι επιδόσεις τους εξαρτώνται από το κατά, έχουν, κατά πόσο κατέχουν καλά την γλώσσα της χώρας υποδοχής. Μετρώντας ε, τις ε, σε σχέση με τις ε, διαδικασίες ε, πίζα αυτές τις επιδόσεις μπορούμε να δούμε το κατά πόσον σε σχέση με την ε, χώρα υποδοχής οι μαθητές που μιλούν μια διαφορετική γλώσσα ποιες είναι οι επιδόσεις τους και βλέπουμε ότι το χάσμα στις επιδόσεις όσον αφορά τις αναλύσεις για τις δεξιότητες ανάγνωσης των δοκιμασιών πίζας, πίζα όταν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι πολλά παιδιά μεταναστών δεν μιλάνε την γλώσσα ε, διδασκαλίας στην οικογένειά τους, στο σπίτι τους. Ένας άλλος τρόπος για να μετρηθεί η επίδοση στη γλώσσα είναι να εξετάσουμε τις επιδόσεις των παιδιών μεταναστών στις δοκιμασίες ψηφιακές ανάγνωσης ε, του, των τεστ PISA. Έχουμε δύο πρακτικά λοιπόν τεστ που ε, εφαρμόζονται όσον αφορά τους υπολογιστές. Η διαφορά είναι ότι χρησιμοποιείται μια πολύ απλούστερη γλώσσα και χρησιμοποιούνται λιγότερα κείμενα σε αυτές τις αναλύσεις. Όμως παρόλα αυτά βλέπουμε ότι οι σχετικές επιδόσεις των παιδιών μεταναστών στις δοκιμασίες ανάγνωσης είναι πολύ χαμηλότερες βλέποντας ε, τις επιδόσεις που είχαν στο πεδίο των μαθηματικών και βλέπουμε ότι οι ακαδημαϊκές ε, ελλείψεις ε, που παρατηρούμε συσχετίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό με την ικανότητα κατανόησης μιας γλώσσας και που ε, κατά τη διάρκεια αυτής της ε, μάθησης διδασκαλίας στο σχολείο μαθαίνουν. Υπάρχει εδώ και ένα δυναμικό των παιδιών αυτών που ε, είναι μεγαλύτερο. Είναι δηλαδή θα, θα λέγαμε μεγαλύτερη η ικανότητα από ότι αυτή που έχει μετρηθεί σε σχέση με την επίλυση προβλημάτων. Δεν είναι όμως όλοι οι μαθητές ε, οι ίδιοι και υπάρχουν διαφορές όσον αφορά την ηλικία άφηξής τους. Ε. Και σε αυτή την ε, καμπύλη βλέπουμε τα παιδιά στο Λουξεμβούργο με διαφορετική προέλευση όταν έχουμε παιδιά που προέρχονται από τη Γαλλία δεν ε, υφίστανται κυρώσεις λόγω της ε, καθυστερημένης άφηξής τους. Άσχετα πότε φτάνουν στο Λουξεμβούργο έχουν σχεδόν τις ίδιες επιδόσεις. Αυτό όμως δεν συμβαίνει με μαθητές από την Πορτογαλία και με μαθητές που προέρχονται από τις χώρες της πρώην Ιουγκοσλαβίας βλέπουμε ότι οι αναλογικές αυτές επιδόσεις, οι σχετικές επιδόσεις ε, ε, φθήνουν σε μεγάλο βαθμό όταν ε, με καθυστέρηση φτάνουν στα σχολεία αυτά τα παιδιά. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να κάνει κανείς ε, λόγο για τις ε, ικανότητες και δεξιότητες της ε, γλωσσικές όταν συζητούμε αυτά τα θέματα. Το να γνωρίζει κάποιος τη γλώσσα της χώρας υποδοχής και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή των κοινοτήτων και να αυξηθεί το αίσθημα ότι ανήκουν κοινωνικά αυτά τα παιδιά σε έναν κοινωνικό περίγυρο. Αυτό το γράφημα δείχνει ότι η πλειοψηφία των παιδιών μεταναστών που συμμετέχουν σε πολιτισμικές δραστηριότητες στις χώρες υποδοχής και βλέπουμε ότι μία μειονότητα ε, χαιρόταν, απολάμβανε αυτή την συμμετοχή. Βλέπουμε λοιπόν ότι το ποσοστό συμμετοχής και το ποσοστό απόλαυσης σε πολύ μεγάλο βαθμό συνδέεται με τις γλωσσικές ικανότητες. Η γλώσσα έχει μεγάλο ρόλο όχι μόνο για την ένταξη των μαθητών αλλά και για την ένταξη των οικογενειών τους στην ευρύτερη κοινωνία διότι είναι μεσολαβητές, διαμεσολαβητές τα παιδιά αυτά μαθητές για τις οικογένειές τους σε σχέση με την κοινωνική τους ένταξη σε σχέση δηλαδή με την κοινωνία υποδοχής και τις οικογένειες προσφύγων που ζουν σε αυτές τις ε, κοινωνίες υποδοχής. Όταν έχουμε λοιπόν το θέμα της ένταξης, τι θα πρέπει να γίνει. Μία σύσταση είναι ότι το εκπαιδευτικό σύστημα θα πρέπει να προσφέρει περισσότερες ε, υπηρεσίες ε, ποιοτικές, αναβαθμισμένες υπηρεσίες ε, μάθησης της γλώσσας όσον αφορά τα παιδιά των μεταναστών. Αυτό το γράφημα δείχνει ότι για τις χώρες και για τις οικονομίες που έχουμε τα στοιχεία 18% των φοιτητών που δεν μιλούν αυτή τη γλώσσα ως μητρική γλώσσα και συμμετέχουν σε τουλάχιστον δύο ώρα μαθήματα ανά εβδομάδα 18% δεν είναι μεγάλο ποσοστό αλλά σε μια μια χώρα σαν τη Σιγκαπούρη είναι 57% αυτό το ποσοστό. Κάτι άλλο που βλέπουμε σε αυτό το γράφημα είναι ότι κάποιες χώρες αναγνώριζαν καλύτερα από άλλες ότι είναι πολυσχηδής διαφορετικός μεταξύ του ο πληθυσμός των μαθητών αλλοδαπών μαθητών ε, από οικογένειες ε, μεταναστών και έτσι λοιπόν ε, όσο το νωρίτερα ξεκινά κανείς τόσο καλύτερα στην Φινλανδία με το παράδειγμα βλέπουμε 32% των μαθητών που δεν είχαν δεν μιλούσαν ως μητρική γλώσσα αυτή, αυτή τη γλώσσα είχαν με, την, με, με με την προσφορά του εκπαιδευτικού συστήματος ε, τις ε, δυνατότητες να προσαρμοστούν καλύτερα. Το ίδιο και για τον Καναδά. Ε, θα ήθελα να αποφύγουμε μια παρανόηση. Κάνουμε λόγο για τη σπουδαιότητα του να υποστηριχθεί η εκμάθηση, μάθηση μιας γλώσσας. Δεν είμαστε υπέρμαχοι μιας πολιτικής που θα έπρεπε μονογλωσσικά καθεστώτα να υποστηρίζει λέμε ότι η εκμάθηση μιας γλώσσας της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι σημαντική υπόθεση αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση για την κοινωνική ένταξη αυτών των μαθητών το να εξακολουθήσουν να έχουν τις δεξιότητες της δικής τους γλώσσας και αυτό γιατί διότι η δική τους γλώσσα βρίσκεται στην καρδιά, στον πυρήνα των παραδόσεών τους και της ταυτότητάς τους και θα πρέπει λοιπόν εδώ σε σχέση με την ταυτότητα της οικογένειας να υποστηριχθεί αυτό το στοιχείο γιατί όταν λένε ότι οι νέοι ε, μπορούν να αποκομίσουν ωφέλη από τις ε, κοινωνίες ε, μέσω αυτής της ένταξης και πάλι κάποιες χώρες περισσότερο από άλλες αναγνωρίζουν ότι η υποστήριξη γλωσσική και με προγράμματα γλωσσικά είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο περίπλοκο από την παροχή απλά και μόνο κάποιων μαθημάτων στην γλώσσα διδασκαλίας της χώρας υποδοχής και έτσι παρέχουν και εκπαίδευση στην ε, γλώσσα, μητρική γλώσσα των παιδιών αυτών, ώστε να μπορούν να ε, διατηρήσουν τις δεξιότητές τους στην γλώσσα τους η αναλογία σε σχέση με αυτό της ε, μιας ε, πολιτικής ε, με ενεργό συμμετοχή στην διγλωσία σε ένα καθεστώς διγλωσίας είναι κάτι που αποβαίνει προς όφελος αυτών των παιδιών. Θα έπρεπε λοιπόν τα σχολεία και τα συστήματα εκπαίδευσης να κάνουν κάτι περισσότερο ώστε τα παιδιά των μεταναστών να μπορέσουν να μάθουν την γλώσσα των σχολείων στα οποία πηγαίνουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής για την ένταξή τους και <clears throat> δεν θα πρέπει μόνο ένα μονογλωσσικό καθεστώς να υποστηρίζεται αλλά ένα ε, πολυγλωσσικό καθεστώς τα στοιχεία μας δεν μπορούν να παράσχουν απαντήσεις σε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, τι είδους δίγλωσης εκπαίδευσης θα ήταν, ε, ε, το καλύτερο και <clears throat> σε σχέση με την διδασκαλία ε, όσον αφορά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα όταν υπάρχει και παράλληλη διδασκαλία της γλώσσας, της μητρικής γλώσσας των παιδιών και σε σχέση με όλες τις ε, δραστηριότητες ε, και πρακτικές ε, που από πλευράς προσωπικού, από πλευράς δασκάλων μπορούν να τύχουν βοήθειας τα παιδιά αυτά ώστε να μπορέσουν να εκτιμήσουν την πολιτισμική πολυμορφία τα παιδιά τα οποία ζουν σε μια βιώνουν αυτή αυτή την κατάσταση στα σχολεία τους. Να δούμε πώς μπορεί δηλαδή η πολιτισμική πολυμορφία από πρόβλημα να αποτελέσει ένα κίνητρο για τη μάθηση, ένα κίνητρο για την προσέγγιση διαφορετικά πολιτισμικών στοιχείων. Ένα φιλόδοξο σχέδιο, ένα φιλόδοξο εγχείρημα έρευνας ε, που βρίσκεται υπό εξέλιξη και συλλέγουμε και στοιχεία σχετικά με αυτό θα δώσει την δυνατότητα να έχουμε περισσότερες απαντήσεις βλέποντας ποια πράγματα έχουν αλλάξει και αλλάζουν ε, αυτή την τελευταία περίοδο σε σχέση με τους μαθητές. Θα προσπαθήσουμε να συλλέξουμε και περισσότερα στοιχεία για να δούμε τι μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι, το διδασκαλικό προσωπικό για να συνδράμουν τους μαθητές μέσα σε, από αυτή την προσπάθεια. Συλλέγοντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία για να μπορέσουμε να δούμε τις ε, προοπτικές των παιδιών αυτών. Σταματώ εδώ και είναι ευπρόσδεκτες οι ερωτήσεις και τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ. Ναι, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ σημαντική σας συνεισφορά. Έχουμε και τις διαφάνειες που ελπίζω να μοιράστηκαν σε όλους. Οπότε θα μπορούμε και στη συνέχεια να μελετήσουμε και να δούμε αυτήν την πανοραμική παρουσίαση της συγκεκριμένης θεώρησης, της γλωσσικής, ε, δια της γλώσσας μάλλον ένταξης και την ένταξη των παιδιών στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα. Και τώρα λόγος στην Μπριζίτ Μπαλκάλμπαχ, Μπάλμπαχ μάλλον, η οποία όπως είπα είναι σχολική διευθύντρια στην, βόρεια, στην νότια σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πρώτα για την πρόσκληση να συμμετάσχουμε και είναι χαρά για αυτό το θέμα το οποίο εξετάζεται σήμερα η δική μας ένωση που το παρακολουθεί και είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το επίπεδο να μπορέσουμε να εκφραστούμε όσον αφορά το προσωπικό στους δασκάλους, ανήκω σε εκείνους που πιστεύουν ότι μια μεγαλύτερη πρόθεση και υποδοχής και ένταξης των παιδιών προσφύγων και μεταναστών αποτελεί συνολική πρόκληση για την Ευρώπη, όχι μόνο για τη Γερμανία από την οποία προέρχομαι και για το ότι όλοι μας από κοινού ακριβώς σήμερα που τόσοι πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες φτάνουν στις χώρες μας πρέπει να συνεργαστούμε αυτά τα παιδιά και οι γονείς τους να μην τραυματιστούν περαιτέρω και να μην αποτελέσουν θύματα ε, της δικής μας, ε, των, δικών μας διαφορών ή αντιπαραθέσεων στην Ευρώπη. Δεν φταίνε γι' αυτό το ότι είναι αλλοδαπή και ότι ήταν θύματα των, ε, της ζωής και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό με ανοιχτό πνεύμα χωρίς να είμαστε προκατηλημένοι από τις πρώτες επαφές με αυτούς τους ανθρώπους όταν περνάνε τα σύνορά μας να δείξουμε τι πρέπει να γίνει. Σας δείχνω, θα σας δείξω ένα παράδειγμα από τη συνεργασία αυτή σε σχέση με το διδασκαλικό προσωπικό κοινωνικούς λειτουργούς ε, υπεύθυνους των σχολείων μας ε, καθώς επίσης ε, και μέλη του κρατηδίου, του, της Βουλής του κρατηδίου μας εργαζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις να μπορέσουμε να επιτελέσουμε αυτούς τους στόχους. Οι δάσκαλοι διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί βρίσκονται στο επίκεντρο, στο σχολείο για την ένταξη αυτών των παιδιών στην κοινωνία μας που με αυτόν τον τρόπο μπορεί η ένταξη αυτή από αυτή την αιστεία από το σχολείο να επιτευχθεί καλύτερα. Γι' αυτό πρέπει οι δάσκαλοι να προετοιμάζονται με τον σωστότερο τρόπο και να βοηθούνται με κάθε τρόπο και γι' αυτό όπως από πλευράς ε, προλαλισάντων... Είμαστε ευγνώμονες για την πρόταση να διπλασιαστούν τα κονδύλια και το, τα μέσα που διατίθενται. Διότι αυτό είναι κάτι στο οποίο χωλένουν οι προσπάθειές μας. Δεν έχουμε το υλικό που χρειάζεται. Οι δάσκαλοι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι όταν μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους και να είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο επιτέλεσης του επαγγέλματός τους. Μαθαίνοντας κιόλας ε, το πώς πρέπει να διδάσκουν γερμανικά ως ε, δεύτερη γλώσσα για αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν με τον καλύτερο τρόπο να έχουν επαφή με αυτά τα παιδιά. Στη Βόρεια Ρινανία αυτό ε, όσον αφορά τις ικανότητες μας ε, και στους δήμους και κοινότητες έχουμε το, τα γερμανικά ως δεύτερη γλώσσα ως μάθημα και, ή τα γερμανικά ως ξένη γλώσσα και έτσι λοιπόν θα πρέπει να μπορούν να εκπαιδεύονται οι δάσκαλοι με αυτόν τον τρόπο τρόπο ώστε να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν προς όφελός τους αυτά τα μαθήματα. Καλό θα ήταν αν είχαμε περισσότερα κονδύλια στη διάθεσή μας. Αυτό διευκολύνει την αντιμετώπιση των προβλημάτων των προσφύγων και των παιδιών, διότι η γλώσσα όπως ακούσαμε διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή τους. Αυτά τα παιδιά δεν, έρχονται μόνο, ή, δεν έχουν μόνο θέματα ε, σωματικά και ψυχικής υγείας, πολλές φορές είναι τραυματικά τραυματισμένα παιδιά, έχουν τραυματιστεί με τα βιώματα τα οποία είχαν. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υποστηριχθούν όπως πρέπει. Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Η δική μας πρόταση είναι να έχουμε πολυεπαγγελματικές μονάδες στις οποίες θα ανήκουν και διερμηνείς, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ήδη στην πρώτη στιγμή υποδοχής ώστε από την πρώτη στιγμή να περιθάλπουν τα παιδιά, να τους παρέχουν εκείνες τις υπηρεσίες, να τα απασχολούν και να παίζουν μαζί μαζί ώστε να υπάρξει συνέχεια στο έργο αυτό της ένταξης. Αυτό μπορεί και με παιχνίδι, όχι υποχρεωτικά μόνο με τη γλώσσα να επιτευχθεί και με θεατρικές ε, ε, παραστάσεις ή δράσεις ε, στις οποίες συμμετέχουν τα παιδιά φυσικά σε μικρές ομάδες. Σημαντικό είναι για μας να μεριμνήσουμε σε αυτό το σημείο αυτά τα παιδιά προσωπικά να αισθάνονται ότι ο ενήλικας απέναντί τους ε, τους απευθύνει τον λόγο για να συμμετάσχουν και να ενεργοποιηθούν έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Θα θέλαμε οι πολυεπαγγελματικές πολυτομεακές ομάδες να μπορέσουν έτσι να εργαστούν και να αλληλοσυνδυάζονται ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των παιδιών. Γι' αυτό θα πρέπει να συνοδεύονται αυτά τα παιδιά στις διάφορες δραστηριότητες ε, της ε, ζωής τους όσο περισσότερο γίνεται ώστε να μπορέσουν ε, οι ικανότητές τους και δεξιότητές τους να αναγνωριστούν έγκαιρα. Έτσι θα διασφαλίζαμε μια συνέχεια στην παροχή περίθαλψης και φροντίδας στα παιδιά αυτά άσχετα σε ποιους απευθύνονται αυτά τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής τους ζωής θα πρέπει να τύχουν αυτής της προσοχής και μέρημνας και να μην αντικαθίσταται αυτό το προσωπικό με διαρκώς άλλους ε, ε, που θα περιθάλπουν αυτά τα παιδιά. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα που θα τους προσφερθεί να επουλωθούν τα τραύματά τους ε, και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να ανακάμψουν και να υπάρξει η δυνατότητα να ε, μπορέσουν να ξεπεράσουν τα όσα βίωσαν. Είναι σημαντικό για τους δασκάλους να μάθουν από ποιο κοινωνικό περίγυρο προέρχονται αυτά τα παιδιά. Καμιά φορά στις τάξεις μας, στα σχολεία μας έχουμε τρεις διαφορετικές γλώσσες οι πέντε διαφορετικές χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μαθητές. Πρέπει να ξέρουν οι δάσκαλοι από ποια χώρα προέρχονται αυτά τα παιδιά, ποια ε, ας το πω έτσι, κοινωνική ένταξη βίωσαν στη χώρα τους υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα κρατήδια μας, στα σχολεία μας, επειδή η θέση της γυναίκας στις χώρες αυτές προέλευσης αυτών των παιδιών και μεταναστών διαφέρει πολύ όσον αφορά τη θέση της γυναίκας στην ίδια τη Γερμανία. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα παιδιά ε, που έχουν ε, τελείως διαφορετικές παραδόσεις ως παιδιά τσιγκάνων ή άλλων που ε, πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη θέση και τον ρόλο της γυναίκας στις κοινωνίες μας. Πρέπει να μπορέσουν οι ε, δάσκαλοι να βοηθηθούν σε αυτό το έργο, να μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν. Δεν ε, ε, θα πρέπει να πούμε ότι επαρκεί το ότι έχουν την επαφή με τα παιδιά. Πρέπει να μπορέσουν να αποκτήσουν τις γνώσεις αυτές για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα παιδιά και οι γνώσεις για τις χώρες προέλευσης είναι σημαντική υπόθεση. Να ξέρουμε τι μπορούμε να τους δώσουμε και τι πρέπει να προσφέρουμε σε αυτά τα παιδιά. Ποια συνέχεια θα δοθεί στα σχολεία, για παράδειγμα στο επίπεδο των ε, ε, κρατηδίων και ε, κοινοτήτων μας πρέπει να έχουμε μια διάγνωση εν που θα διαπιστώνει ποια είναι η σωστή θέση ποιου παιδιού σε ποιο σχολείο ώστε να έχουμε τους σωστούς δασκάλους απέναντί τους. Στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία στο ε, κοινοτικό επίπεδο ε, διασφαλίζεται αυτή η υπηρεσία διότι έχουμε σε σχέση με τους ε, πρόσφυγες ξεχωριστές ιδιομορφίες που πρέπει με επαφή με τους γονείς με μια πρώτη αξιολόγηση να μπορέσουμε να διαγνώσουμε ποια είναι η κατάσταση των παιδιών ποια είναι η ιδιομορφία των καταστάσεων αυτών ώστε να μπορέσουμε με βελτιωμένο τρόπο να εργαστούμε. Μπορούμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό μέσω της μακράς παρατήρησης ε, παιδιών. Πρέπει με συστηματικό τρόπο να γίνεται αυτό και όχι μόνο με, μια, ε, ένα ρηχό τρόπο βιαστικά ή με μια πρώτη ματιά. Θα πρέπει με καταλόγους ε, που πρέπει να ε, συμπληρώσουν στοιχεία δάσκαλοι για τα παιδιά αυτά με την παρατήρησή τους μέσα από ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με τα παιχνίδια, με τα αθλήματα, με τις πολιτιστικές δραστηριότητες, με τα βιώματα των παιδιών, να αφήνουμε χώρο για το παιχνίδι, χώρο, και χρόνο για το παιχνίδι των παιδιών. Είμαι υπέρ, για παράδειγμα, του ότι οι πλοηγή οι πιλότοι ένταξης που σε αυτούς θα ανήκουν και διερμηνείς ε, με δεξιότητες ε, να μπορέσουν ε, γνωρίζοντας τις ανάγκες των παιδιών να είναι οι σωστοί διαμεσολαβητές γνωρίζοντας τα παιδιά και τις ανάγκες τους και εδώ να μπορούν να εξηγήσουν στα παιδιά το τι είναι το ένα είναι το άλλο ή άλλο πράγμα παρόλα αυτά θα υπάρξει η εγγύηση μέσω αυτής της προσέγγισης ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, ένταξη αυτών των παιδιών με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Στενή επαφή με τις οικογένειες, ε, το ανέφερα αυτό και μπορούμε επαγγελματικά να παράσχουμε και βοήθεια. Δεν έχουν επιτευχθεί όλα αυτά, δεν είναι όλα δεδομένα, εργαζόμαστε για να τα πετύχουμε. Τα γερμανικά ως ε, δεύτερη γλώσσα θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό μάθημα για αυτά τα παιδιά. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες τάσεις που λένε πρέπει να βάλουμε τα παιδιά σε σε μια ε, συγκεκριμένη ε, γερμανική τάξη για να ενταχθούν σε αυτήν. Δεν είναι αυτό το πιο αποτελεσματικό. Ε, τα παιδιά αυτά που αισθάνονται μεγάλη πίεση πρέπει να μπορέσουν με τη γλώσσα που θα μάθουν, τη γλώσσα της, τη γερμανική γλώσσα, να μπορέσουν να προχωρήσουν αν κάποιος ε, δεν γνωρίζει την, δεν έχει μάθει τη γλώσσα όπως θα έπρεπε, τότε δεν μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσεις, δεν μπορεί να εκφραστεί και να επικοινωνήσει και αν θέλουμε να υπάρξει πραγματική σωστή προσφορά αντικειμένων στην, ε, στο σχολείο, δηλαδή μαθημάτων που θα πρέπει να μπορούν να αφομοιώσουν τα παιδιά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μάθουν πρώτα τη γλώσσα για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μετά και θα πρέπει εδώ να δούμε τις, ε, τα, τα ε, κενά που υπάρχουν. Αν δεν τα καλύψουμε ευθύ εξ αρχής θα συνεχίσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής του ζωής ε, να έχουν αυτές τις ελλείψεις τα παιδιά και δεν θα μπορέσουν ποτέ να εκμεταλλευτούν το πλήρες δυναμικό τους. Ε, σπάνια υπάρχουν τάξεις παιδιών που, είναι, που αποτελούνται συναπαρτίζονται μόνο από παιδιά ε, μεταναστών. Έτσι λοιπόν στην ε, Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία υπάρχει η πολιτι, πολυπολιτισμική ε, τάξη ας το πω έτσι όπου σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ε, παιδιά ε, που έχουν ενταχθεί σε αυτές τις τάξεις έχουν και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ τους πρόκειται για την ποιότητα των μαθημάτων που παρέχεται και να δούμε το κατά πόσον τα παιδιά μπορούν πραγματικά να αποδώσουν. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα οποία εμείς προσπαθούμε προσπαθούμε να τους μάθουμε μπορούν και τα παιδιά να αφομοιώσουν και να τα μάθουν. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει ένταξη. Και έχουμε κάθε συμφέρον λοιπόν σε μια τάξη που υπάρχουν παιδιά μεταναστών να μπορέσουμε να τα βοηθήσουμε να μην έχουν και να ε, στα όσα έχουν θα έπρεπε να είχαν μάθει. Για να μπορέσουμε την κοινωνικοποίηση των παιδιών αυτών και την ένταξή τους ε, στις ε, κοινωνίες μας να την επιτύχουμε και των οικογενειών τους κιόλας και εμείς πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, να ε, μάθουμε να τους εκτιμάμε και να τους ε, προσεγγίσουμε σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο τώρα να προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο τι πρέπει να γίνει για, τους, για τις οικογένειές τους και οι γονείς αυτών των παιδιών οι οικογένειές τους πρέπει να τύχουν αυτή της προεργασίας για να μπορέσουν να συνεννοούν και ε, με, την κοινωνία και τους καθηγητές να αναγνωριστούν ε, τα, οι ελλείψεις και τα κενά να μπορέσουμε την βούληση που πρέπει να υπάρχει από πλευρά των γονέων και των παιδιών να την εντάξουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην κοινωνικοποίησή τους. Πρέπει εμείς οι δάσκαλοι να προετοιμαστούμε για αυτή τη διαφορετική προέλευση αυτών των παιδιών και τη διαφορετικότητα των γονιών τους και των οικογενειών τους. Σημαντικό θα ήταν σε κοινέ δραστηριότητε ε, σε ε, τέτοιε α το πω επαφές ε, γονέων να προχωρήσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε δραστηριότητε για την κοινωνική ένταξη που θα είναι σημαντικές, να μπορέσουμε για παράδειγμα να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα μάθησης ή σχολικής επίδοσης των παιδιών. Υπάρχουν διαφορετικές δραστηριότητες ε, που θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε κάποιες προτάσεις που έχουμε υποβάλει στο Υπουργείο μας και ελπίζουμε ότι κάτι θα γίνει στο τέλος τέλος. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε μια ολόκληρη αλυσίδα εκπαίδευσης και προετοιμασίας που όχι μόνο στα σχολεία αλλά και με άλλες πολιτιστικές δράσεις ε, πρέπει να συνοδεύεται και να δένει εκ παραλίλου ώστε μακροπρόθεσμα όλο και μεγαλύτερη τεχνογνωσία να μπορεί να ε, επενδύεται σε αυτές τις δράσεις. Αλλά όχι μόνο σε εμά, αλλά και στα άλλα κρατήδια της Γερμανίας και παντού στην Ευρώπη θα πρέπει υπερπεριφερειακά πέρα από κρατικό επίπεδο να επενδύσουμε σε αυτές τις δράσεις. Και εδώ προτείνουμε ένα συγχρονισμό που θα βοηθήσει στο να ε, διευκολυνθεί το έργο μας ε, ευρωπαϊκά και να μπορεί όταν κάποιος ε, μετακινείται κάπου αλλού να μπορεί να έχει κάτι το αντίστοιχο, κάτι παράλληλο μέσα σε μια συνολική προσέγγιση, σφαιρική προσέγγιση σε διαφορετικά επίπεδα. Σήμερα μέσω του σχολείου μέσω της κοινότητας, μέσω της περιφέρειας, υπερπεριφερειακά στο κρατήδιο, στην όλη σε, στο ε, εθνικό επίπεδο θα μπορούμε να δράσουμε και θα μπορέσουμε έτσι να και ολοκληρώνω το έργο της κοινωνικής ένταξης ε, να το εντάξουμε και στο, ε, στον στόχο και στις πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε για την εκπαίδευση. Εκπαίδευση και δασκάλων και επικουρικά επαγγέλματα ή και νέα επαγγέλματα τα οποία θα εντάξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας και να σκεφτούμε ότι πολυεπαγγελματικές, πολυτομεακές τέτοιες ομάδες θα ήταν μια δυνατότητα που θα έδινε την δυνατότητα στο το δυναμικό που έχουμε να το ενδυναμώσουμε και να το εκμεταλλευτούμε καλύτερα. Θα πρέπει με καινοτόμο τρόπο να σκεφτόμαστε, με νέες ιδέες να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων ακόμα και αν υπάρχει μία ιδέα είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι να μην ε, ε, υπάρξει τέτοια κατάσταση που να ξεπερνά τις δυνατότητες και ικανότητές μας. Πολλές φορές ε, ξεπερνά τις δυνατότητες ενός δασκάλου όταν δεν υπάρχει το υλικό το οποίο χρειάζεται ή η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάλμπαχ. Ήταν σημαντικό να ακούσουμε τις απόψεις μιας εκπαιδευτικού, ε, διευθύντριας μάλιστα, με τόσο σημαντική πείρα για ένα τόσο σφαιρικό πρόβλημα, αυτό των δασκάλων στην Ευρώπη. Έχουμε καθυστερήσει βεβαίως κάμποσο, οπότε Θα έλεγα να περάσουμε στις ερωταπαντήσεις σε αυτή τη φάση, αλλά πολύ γρήγορα, ένα λεπτό ο καθένας, όποιος θέλει να κάνει μια ερώτηση, και να προσπαθήσουμε να είμαστε σύντομοι και στις απαντήσεις, γιατί έχουμε άλλα δύο πάνελ. Η σειρά με την οποία γράφησαν στον κατάλογο αγορητών οι ομιλητές. Φερχάιεν, Λιμπάτσκα και μετά συνεχίζουμε. Δύο σύντομες ερωτήσεις συγκεκριμένα όσον αφορά την, ε, την διδασκαλία της μητρικής γλώσσας ε, που θα πρέπει να παρέχεται. Ακούσαμε από πλευράς εκπροσώπου του ΩΣΑ ότι οι ικανότητες στη μητρική, ρόλο, στη μητρική γλώσσα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και σε σχέση με την γλώσσα της χώρας υποδοχής και πρέπει εδώ παράλληλα να υπάρχει εκμάθηση ή καλλιέργεια της, και των δύο γλωσσών ώστε στη γλωσσική δομή που θα παρέχεται να αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της διαφορετικής γλώσσας που ομιλείται στην οικογένεια του παιδιού από τη γλώσσα που ομιλείται στο σχολείο και θα πρέπει να υπάρχει επαρκής δομή γλωσσική με την ε, ε, ε, βοήθεια που θα παρέχουμε στα παιδιά αυτά διτά. Αυτό είναι ερώτημα τώρα προς εμάς κύριε γίνεται αυτό, πόσο μπορεί αυτό να αντιμετωπιστεί. Και η δεύτερη ερώτηση προς ε, την κυρία Προλαλή Είχαμε μια παρόμοια κατάσταση όταν είχαμε πρόσφυγες από την Ανατολική Ευρώπη, κυρίως από τη Ρωσία, που είχαν έρθει σε εμά με παιδιά διαφορετικών ηλικιών και είχαμε παράλληλες τάξεις που είχαν δημιουργηθεί στα σχολεία μας και υπό το πρίσμα είναι καλύτερο λέει, να μαθαίνουν τα παιδιά στη, τη μητρική γλώσσα, τη, να συγχωρείτε τη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Εσείς λέτε ότι πρέπει να υπάρξει η, ε, ε, ε, υποβοηθητικός που θα δίνεται σε αυτά τα παιδιά για να μαθαίνουν και τη δική τους γλώσσα. Πώς μπορούν λοιπόν παιδιά μεταναστών με διαφορετικές γλώσσες, πώς αυτές θα διαφοροποιούνται όσον αφορά μια τέτοια τάξη μαθημάτων και παιδιά που έχουν τα αραβικά ως μητρική τους γλώσσα με παιδιά για παράδειγμα από το Αφγανιστάν όταν βρίσκονται σε μία τάξη πώς αυτό το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσει Ευχαριστώ πιο γρήγορα μπορείτε να γιατί δεν θα προλάβουμε Λιμπάτσχα και μετά Σφέρ Ευχαριστώ πολύ Εμείς ακούσαμε δύο πραγματικά ενδιαφέροντα σημεία Καταρχήν ε, αναφερθήκατε στο ότι υπάρχουν ενώσεις όπως αυτή της ε, ε, αυτή των Ρωμά όπου οι Ρωμά δεν θέλουν να συμμετέχουν σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα όπου δεν υπάρχουν δάσκαλοι Ρωμά και δεν καταλαβαίνω και αυτό σας ρωτώ, πώς μπορεί να εκπαιδεύσει κανείς δασκάλους με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο όταν ανήκουν σε άλλη γλώσσα. Δηλαδή είναι διαβίου εκπαίδευση, είναι κάτι διαφορετικό. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το γεγονός πως η ενσωμάτωση βοηθά στο να ανοίξει μια κοινωνία είναι ε, μια βασική παραδοχή και αποτελεί και στόχο εδώ και πολλά χρόνια γιατί στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ακριβώς την ενσωμάτωση. Το να κλείνουμε τους ξένους μέσα σε γκέτο βεβαίως και δεν είναι το κατάλληλο. Οπότε χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση έτσι ώστε οι πρόσφυγες να ενσωματώνονται. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά γιατί τα παιδιά μπορούν να συνεισφέρουν πάρα πολλά στην ενσωμάτωση γιατί βοηθάνε και τις ίδιες τους τις οικογένειες και διευκολύνουν την επικοινωνία μέσα σε καταστάσεις στις κοινωνικές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους, δηλαδή όταν πάει οικογένεια στο γιατρό κτλ. Οπότε σας έδωσα ένα πρακτικό παράδειγμα του ποιος είναι ο ρόλος του παιδιού σε αυτή την περίπτωση. Η παρέμβαση που ακούσαμε για το θέμα της κρίσης της ε, κοινωνικής ένταξης και για το γεγονές πως υπάρχουν πολιτισμικά μοντέλα πολύ διαφορετικά μέσα στην ίδια κοινωνία, σήμερα μας έχει οδηγήσει ε, σε ένα είδος προσπάθειας ε, για ιδεολογική ε, ένταξη, δηλαδή να μπορούμε να δεχόμαστε τα κοινωνικά μοντέλα αλλήλων και δεν ξέρω αν οι Ευρωπαίοι είναι ακόμα έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Ο κύριος Ταρτζεντίνη έχει το λόγο με συγχωρείτε, ε, στον κύριο Αργεντίνη θέλω να κάνω την ε, ερώτηση αυτή, γιατί μιλώ, μιλήσατε για παιδιά ε, τα οποία σε κάποια σχολικά συστήματα ενσωματώνται πιο πετυχημένα, είναι πιο αποδοτικά, ενώ σε άλλα όχι. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι έκανε η συγκεκριμένη χώρα για να δίνει την αίσθηση αυτή του ανήκειν στους μαθητές, έτσι ώστε αυτοί με τη σειρά τους να αποδίδουν καλύτερα. Η κυρία Κινίτσι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τις παρουσιάσεις που ακούσαμε και να καταγράψω την πραγματική ανάγκη στην πράξη να διοργανωθούν δράσεις ένταξης για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις περιθωριοποίησης τις οποίες είμαστε μάρτυρες όλοι σήμερα. Μια ερώτηση βάσει μιας προσωπικής μου εμπειρίας ε, στη δουλειά μου. Ε, ήμουν ε, εισαγγελέα για τους ανηλίκους εισαγγελέα στην Ιταλική Δημοκρατία επί σειρά ετών και ξέρω πολύ καλά ότι υπήρχαν θέματα με ανηλίκους άλλο δαπούς, ελάχιστους ε, ομολογουμένως, που ήταν σε κράτηση σε κάποιες από τις δικές μας εγκαταστάσεις και δομές. Προκειμένου να βοηθήσουμε τους αλλοδαπούς ανηλίκους να ενταχθούν μαζί με τους πολιτιστικούς διαμεσολαβητές θα έπρεπε να πειραματιστούμε και με την ιδέα οι ανήλικοι της Ιταλίας να ασχοληθούν με αυτή τη διαδικασία ένταξης και να το συνοδεύσουν. Ακριβώς για να ενισχυθεί το αίσθημα του ανήκειν με μία γλώσσα ισότητας που μπορούν να μιλήσουν οι νέοι μεταξύ τους, ε, νέα παιδιά που μπορούν να καταλάβουν την κατάσταση των άλλων νέων παιδιών, ε, ακόμη και αν είναι πρόσφυγες, αυτό μπορεί να τους βοηθήσει να ενταχθούν με μία χείρα βοηθείας που έρχεται από τα ίδια τα παιδιά. Εδώ λοιπόν είχαμε ως τώρα εμείς στην Ιταλία πολύ θετικές εμπειρίες. Ε, ρωτώ λοιπόν θα μπορούσαμε με τις απαραίτητες προσαρμογές να σκεφτούμε κάτι τέτοιο, να υπήρχε ένα τέτοιο εγχείρημα και για τα σχολεία. Αυτό το ερώτημα ήθελα να θέσω στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Κατερίνα. Ο κύριος Νέκοφ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και θα είμαι και πολύ σύντομος, γιατί ξέρω πως δεν υπάρχει χρόνος. Όπως είπε πολύ σωστά και ο κύριος Σιέρ, τα παιδιά ε, θέλουν να προχωρήσουν. Και όταν θέλουν να προχωρήσουν βοηθάνε και τους γονείς να ενσωματωθούν πιο γρήγορα. Τι κάνουμε όμως με την περίπτωση των παιδιών που αρνούνται να ενσωματωθούν. Εδώ κάνω μια σύγκριση μεταξύ των ε, παιδιών που τα παιδιά που ε, βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, εκτός απασχόλησης. Αν δεν θέλουν να ενσωματωθούν λοιπόν μπορούμε να τα απομακρύνουν από τις κλειστές κοινωνίες μέσα στα οποία εγκλωβίζονται και έτσι δεν θέλουμε να ενσωματωθούν γιατί διαφορετικά θα μετακινηθούν προς το περιθωριοποιημένο κομμάτι της κοινωνίας όπως για, συμβαίνει με τα παιδιά τα οποία είναι εκτός, εκ, εκτός παιδείας, εκτός απασχόλησης, εκτός εργασίας, τα νίτς δηλαδή. Νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τις περιθωριοποιήσεις περισσότερο από οτιδήποτε κάτι άλλο, όπως επίσης και από την ριζοστικοποίηση. Και τρία λεπτά στον καθένα για τις απαντήσεις σας. Παρακαλώ πολύ να ξεκινήσουμε με τον κύριο Πιατσεντίνη για το θέμα το κατά πόσο είναι πρόβλημα το ότι μιλάνε διαφορετικές γλώσσες στο σπίτι ε, οι μαθητές σε σχέση με τη γλώσσα στην οποία μαθαίνουν στο σχολείο δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα ε, η διγλωσία είναι απόλυτα εφικτή για τους περισσότερους μαθητές και όχι μόνο από τους μαθητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ νέοι, αλλά και από παιδιά τα οποία είναι στα 10-15. Όπως επίσης αποδεικνύεται πως το να αποκτήσει κανείς Ε, ικανότητες ε, αρκετές σε μια τρίτη ξένη γλώσσα ε, είναι απόλυτα αφικτό και πάλι για τους περισσότερους. Είναι δηλαδή μια γνωστική ικανότητα που αναπτύσσεται σε όλους. Μπορούν τα παιδιά, ε, να μιλάνε με τους συμμαθητές σε άλλη γλώσσα και άλλη γλώσσα στο σπίτι. Δεν χρειάζεται να ζητάμε από τους γονείς να μιλάνε ε, στη γλώσσα της χώρας υποδοχής. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις τελικά αυτό απλώς ε, μειώνει την ενσωμάτωση του ατόμου και δημιουργεί οικογενειακά προβλήματα. Τώρα για την διαφορά που έχουμε σε, μεταξύ κρατών, ναι, είναι διάφοροι όμως οι παράγοντες και δεν είναι μόνο τα σχολεία, έχει να κάνει με τα σχολεία και τις κοινωνικές πολιτικές που ακολουθούν γιατί ένας βασικός λόγος που δημιουργεί αυτή την αίσθηση του ότι ανήκει ή όχι είναι τι κάνεις με φτωχούς ε, μαθητές οι οποίοι ζουν σε περιο, περιοθωροποιημένες ε, ε, ομάδες κοινωνικές, κατά πόσο δηλαδή το κοινωνικό κράτος πρόνοιας τους βοηθά έτσι ώστε να ξεπεράσουν αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις φτωχές κοινωνίες. Και αυτό μας το ε, εξηγεί καλύτερη περίπτωση της Φιλανδίας, δηλαδή το τι μπορούν να κάνουν οι δάσκαλοι, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα εργαλεία για την ε, γρήγορη αναγνώριση των γλωσσικών δυσκολιών, όπως επίσης και του θέματος της επιμόρφωσης των δασκάλων. Αλλά είναι ένα μεγαλύτερο θέμα, το οποίο έχει να κάνει ε, με την ε, υπερπίδηση των εμποδίων. Τώρα το peer learning, το μαθαίνει κανείς δηλαδή από τους ε, ε, όσου είναι γύρω τους, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί πολύ με τα παιδιά και τα στοιχεία που έχουμε και που συνδυάζονται με τις δραστηριότητες στην τάξη, μέσα, με, την, με τον πολιτισμικού χαρακτήρα και τις ε, διαφορές που ε, βλέπονται, που αναγνωρίζονται ως πλούτος μέσα από το μαθητικό σύνολο. Τώρα για το άλλο θέμα που αναφέρατε, νομίζω ότι είναι πολύ λίγοι οι μαθητές οι οποίοι δεν θέλουν ε, να ενταχθούν. τα παιδιά θέλουν αντίθετα την αναγνώριση των συνομιλίκων τους, οπότε νομίζω ότι δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό ως πτυχή. Ich hoffe, ich bin zu hören. Ja, danke. Ακούτε, ελπίζω. Ναι. Τώρα, την κανονική τάξη ή τις, ε, τα γλωσσικά μαθήματα. Πιστεύω ότι από τα όσα έχω ακούσει από συναδέλφους μου, Χθε ε, είχα και καθηγητές από διάφορα σχολεία και ρώτησα τι θα συνιστούσατε. Θα ακολουθούσατε αυτά δηλαδή τα οποία εγώ σας εξέθεσα ή θα λέγατε καλύτερα όχι. Και είπαν με σαφήνεια ότι είναι υπέρ τουλάχιστον ένα εξάμεινο πιο πριν να γίνεται αυτό. Όχι δηλαδή με τους άλλους να μην ακολουθούμε τέτοιες δραστηριότητες. αντίστροφα έδωσαν και παραδείγματα όταν πάνε στραβά τα πράγματα σε μια τάξη γιατί δεν καταλαβαίνουν κάποια παιδιά κάποια πράγματα υπάρχουν ευθύ εξ αρχής από τη ε, σχολική τους ε, σταδιοδρομία κενά και ελλείψεις και αισθάνονται άσχημα. Θέλουν να μπορούν να συμμετάσχουν και να μην περιθωριοποιούνται και νομίζω ότι αυτό θα απάμπλυνε την κατάσταση αν είχαμε ένα τέτοιο πρότυπο και προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά έτσι. Προσπαθούμε να τα καταφέρουμε. Σημείωσα εδώ ποια είναι τα προσωπικά βιώματα με τις ομάδες. Ναι, αλλά δεν έχουμε ακόμα τέτοιες ομάδες. Όλα τα κάνουμε μόνοι μας στη, στη Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία. Εμείς θα πρέπει να δώσουμε, ε, κάνουμε και ενέσεις καμιά φορά όταν κάποιος είναι άρρωστος και πρέπει όλα αυτά να μας βοηθήσουν από πλευράς της υπηρεσίας μας. Σας λέω πώς έχουν τα πράγματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει πίεση πρέπει να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτές τις ικανότητες, αυτές τις δεξιότητες, πρέπει να έχουμε περισσότερο ευρύτερο φάσμα ε, δραστηριοτήτων αλλά μας αφήνουν μόνους μας, αβοήθητους ε, και δεν υπάρχει και επιμόρφωση ή εξειδίκευση. Για παράδειγμα για την διδασκαλία γερμανικών ως ξένης γλώσσας. Ε, και εδώ από πλευράς του Υπουργείου με τους όσους έχουν στείλει ζήτησα απίθυνα αίτημα οι συνάδελφοί μου στις, ε, στις τάξεις που έχουν ε, των παιδιών να μπορούν να εκπαιδεύονται όπως πρέπει. Δεν έχουμε όμως αυτή τη δυνατότητα και μπορείτε να φανταστείτε ποια απογοήτευση νιώθουν αυτοί οι δάσκαλοι όταν δεν μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί όπως πρέπει. <clears throat> Δεν έχουμε χρήματα όπως θα έπρεπε να είχαμε, δεν έχουμε επαρκή κονδύλια. Μετά σημείωσα εδώ κάτι άλλο. Α, επιμόρφωση, περαιτέρω κατάρτιση, εντάξει το ανέφερα. Αλλά ε, επίσης ε, έχω ε, σημειώσει εδώ τις ε, δεξιότητες. Ας το πω εξής. Η προλαλή σας είπε κάτι καταπληκτικό. Πρέπει την αλληλεγγύη να εκφράζουμε να εκφράζεται η αλληλεγγύη και πέρα από τις επιφυλάξεις που μπορεί κανείς να έχει να ξεπερνά τους δισταγμούς και τις επιφυλάξεις του και εγωισμός όπως αναφέρθηκε να ξεπερνάμε τις εγωιστικές τάσεις ναι, αλλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι εγωιστές. Δεν είναι ο εγωισμός που πρέπει να ξεπεράσουμε. Οι φοβίες μας και οι φόβοι μας είναι αυτό που πρέπει να ξεπεράσουμε. Πολλοί, πολλές φορές φοβούνται την αλλαγή ή κάτι καινούριο ή άγνωστο. Μπορώ να σας πω σε σχέση με τη Γερμανία, αν εμείς τις αξίες μας, τις χριστιανικές αρχές και αξίες και όταν έχουμε και ανθρωπιστικές αξίες, αν εμείς γνωρίζαμε αυτές τις αξίες όπως και οι μουσουλμάνοι έχουν εξοικειωθεί με τις δικές τους αξίες, ε, δεν θα χρειαζόταν να έχουμε φοβίες και φόβους. Σας ευχαριστούμε για αυτό το συμπέρασμα. Νομίζω ότι πραγματικά αυτή η έκκληση των δασκάλων αφορά όλους τους δασκάλους στην Ευρώπη και πραγματικά Θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μα προ του δασκάλου τη Ευρώπη. Γιατί πολύ συχνά είναι στην πρώτη γραμμή, στην εμπροστοφυλακή τη υποδοχή. Και πολλέ φορέ το σχολείο με τις βέλτιστες πρακτικέ που υπάρχουν, όσο φανταστικέ κι αν είναι, ε, δεν γίνεται γνωστό. Ε, δεν γίνονται γνωστέ οι δράσει στα σχολεία. Ε, ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Δόκτωρο Πιατσεντίνη. Και τώρα πολύ γρήγορα να περάσουμε στους επόμενους εμπειρογνωμονές μας. Αλλάζει το πάνελ. θα τους υποδεχτούμε τόσο λίγο και αν θέλετε κι εσείς κύριε για να λάβετε το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ακούσουμε την κυρία Μέλανη Ήμπελ Uh, Καλώ την κυρία Μελανίμπελ του Συμβουλίου Νέων του Βραδεμβούργου. Παρακαλώ. Έπειτα η κυρία Έλενα Μπεζότσι της Επιστημονικής Επιτροπής του Παγκόσμιου Ιδρύματος Μεταναστών στη Ρώμη. την. Και μετά οι κυρίες κυρίες Μαριάν Πονσλέ και Πατρίς Βίτσερφ. του Διεθνούς Ιδρύματος ε, Γεχοντήμενου Χιν στο Βέλγιο. Έχουμε λιγότερο χρόνο από ό,τι προβλεπόταν, οπότε θα σας παρακαλέσω όλες να είστε, εάν γίνεται, συνοπτικές στις παρουσιάσεις σας. Πάντως είναι χαρά μου που βρίσκεστε εδώ και ε, κύριε Καριάτσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προϊσταμένη της υπηρεσίας για το πρόγραμμα Εράσμους. Και όλο όλες τις υπηρεσίες και για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της Ευρώπης του 2020 και για το Erasmus πλάσου. Να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στην κυρία Μέλανη Ήμπελ από το Συμβούλιο των Νέων. Παρακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα αυτή μέσα στο πλαίσιο αυτής της ακρόασης να τοποθετηθώ για την εμβέλεια της πολιτικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης, εκπαίδευσης και μέσα σε έναν άτυπο και σε ένα άτυπο πλαίσιο. Ονομάζομαι Μελανή Έμπερ και εργάζομαι στο Συμβούλιο Νέων του Βραδενβούργου. Είμαστε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Νέων και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων που εκπροσωπούμαστε εδώ. Το κρατήδιο Μπραντεμπορ που ανήκει στην πρώην Ανατολική Γερμανία το 2015 είχε περίπου 28.000 ε, πρόσφυγες που ε, δέχτηκε σε αυτό. Το 2016 άλλοι 40.000 αναμένονται να προσέλθουν σε εμά. Τουλάχιστον 30% από αυτούς όλους είναι παιδιά και νέοι κάτω από 18 ετών Κατά το προηγούμενο καλοκαίρι χαρακτηρίστηκε η Γερμανία από ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης και προθυμίας Γερμανών να βοηθήσουν μέσα στο πλαίσιο των καλοδεχούμενων εντός εισαγωγικά αυτών ε, πληθυσμών και των νέων. Τώρα, λίγο αργότερα, έχουμε την κατάσταση όπου έχουμε μια διαφορετική εικόνα πλέον. Υπάρχει η εχθρότητα προς τους ξένους που έχει αυξηθεί και μάλιστα έντονα. Μια εικόνα που από την προηγούμενη κυρία Κυριακή εδώ και τρεις ημέρες μέσω της αύξησης ε, των μεταεκλογικά αποτελέσματα που σημειώθηκαν της ΑΕΦΔ της εναλλακτικής δηλαδή λίστας της Γερμανίας, ε, μας δείχνει τι συμβαίνει. Είναι έργο μας ε, σε περιφερειακό, τοπικό και εθνικό επίπεδο αυτό το κύμα, το ξενοφοβικό και το εχθρικό προς τους ξένους, να το αντιμετωπίσουμε με τοπικά, με μια φιλική προς τους ξένους στάση και τοποθέτηση. Και πρέπει να δούμε τα μέτρα σε σχέση με την Επιτροπή, Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών όπως προτάθηκαν και πρέπει και αναφέρθηκε αυτό να είμαστε πρόθυμοι να αλλάξουμε και να βοηθήσουμε στην ένταξη αυτών των ε, ε, ανθρώπων και να διασφαλίσουμε για τους νέους αυτούς κατοίκους του κρατηδίου μας παράλληλα με τους παλαιότερους μια θετική συμβίωση. Αυτό θα έχει σημαντικό ρόλο κατά το επόμενο διάστημα για την ένταξη αυτών των ανθρώπων ανθρώπων. Χρειαζόμαστε τη σωστή προσέγγιση σε μια περίοδο κρίσης όπου η εκπαίδευση, η παιδεία, η δημοκρατία θα είναι οι κυριότερες έννοιες ώστε αφενός οι νέοι αυτοί πολίτες να αποκτήσουν προοπτικές στη ζωή τους και από την άλλη πλευρά να ενισχυθεί η δημοκρατική τάξη πραγμάτων στη χώρα μας. Η πολιτική και πολιτιστική εκπαίδευση συνεισφέρει σημαντικά προς αυτό το στόχο. Η συζήτηση για την αξία της άτυπης εκπαίδευσης εκτός, σχολείων από τη μελέτη που συντάχθηκε, μελέτη πίζας όπως την αποκαλούμε το 2000 έχει όλο και μεγαλύτερο ρόλο που αποκτά. Ένας ένα μεγάλο τμήμα της άτυπης αυτής ε, παιδείας και εκπαίδευσης ε, από τη δεκαετία του 70 ε, καλύπτουν τα Συμβούλια Νέων σε εταιρική σχέση με εργαστήρια για τους νέους και πολλές πολλές άλλες μονάδες και φορείς συμμετέχουμε σε αυτό, στην επιτέλεση αυτού του στόχου. Σε εταιρική σχέση με τα κρατικά όργανα και φορείς και μέσα από μια δράση ανεξάρτητη να μπορέσουμε να προσφέρουμε ως Συμβούλια Νέων στα παιδιά και στους νέους τη δυνατότητα να συμμετέχουν μέσα σε ένα πλαίσιο επομισμού ευθύνη να ζήσουν την δραστηριοποίησή τους και τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριοποίησής τους κοινωνικά να μπορέσουν να διαμορφώνουν δικούς τους χώρους δράσης και να αποκτούν τις αναγκαίες δεξιότητες και ικανότητες για να τα βγάλουν πέρα στη ζωή τους οι πολύμορφες προσφορές σας ε, σε αυτούς τους νέους εξυπηρετούν το να βοηθηθούν αυτοί οι νέοι να ενηλικιωθούν, να ε, ανεξαρτοποιηθούν, να υλοποιήσουν τα όνειρά τους και τις αξίες τους και έτσι να ενισχυθεί η ίδια η δημοκρατία και να προαχθεί το δημοκρατικό καθεστώς. Με την προσέγγιση των, της εμπειρικής ε, εργασίας και της, του σεβασμού των δικών τους προτεραιοτήτων θα πρέπει με σεβασμό της πολυμορφίας ε, να πούμε ότι τα Συμβούλια Νέων δραστηριοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια συνεισφέροντας σημαντικά για την ε, ένταξη και ε, αυτοεκπλήρωση των στόχων αυτών των επιθυμών, επιθυμιών αυτών των νέων. Λαμβάνοντας τώρα υπόψη εδώ και τις ανάγκες των νέων που είναι πλέον παιδιά μεταναστών χωρίς να υπάρξει καμία στιγματοποίηση ή περιθωριοποίησή τους. Θα πρέπει να βοηθήσουμε βοηθήσουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά των προσφύγων και μεταναστών. Υπάρχει, ε, πολυάριθμη, υπάρχει ευρύ ε, φάσμα εμπειριών με ειδικού χώρους που μπορούμε να διαθέσουμε στα παιδιά αυτά των Συμβουλίων Νέων ή των ε, ε ας το πω κέντρων νέων ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν τα παιδιά αυτά το ένα το άλλο οι δυνατότητες αθλημάτων και ελεύθερου χρόνου ώστε να μπορούν να να συμμετάσχουν τα παιδιά προσφύγων ε, δραστηριότητες καλλιτεχνικές, ε, μουσικές, ε, θεατρικών παραστάσεων και δραστηριοτήτων που πολιτιστικά θα μπορέσουν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά και να ξεπεράσουν τον γλωσσικό φραγμό για να μπορέσουν να συμμετάσχουν μέχρι και εξειδικευμένα σεμινάρια για παιδιά προσφύγων και πρόσφυγες ώστε να εξοικειωθούν με το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας και να τους εξηγήσουμε πώς έχουν τα θρησκευτικά θέματα και κοινωνικά θέματα στη χώρα μας ιδιαίτερα καλά μπορούν να πετύχουν τα προγράμματα σε περιοχές όπου έχουν ήδη προηγούμενη πείρα και εμπειρία ε, σε περιοχές μας σε αντίθεση με τη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία στο Βρανδεμβούργο είχαμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό αλλοδαπών 2,6% επίσης πολύ χαμηλό ποσοστό σε σχέση και με άλλα ανατολικοευρωπαϊκά κρατήδια υπήρχε πολύ στενό πλαίσιο επαφών ε, με αλλοδαπούς δεν είχαν τέτοιες επαφές και δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ε, τη διαφορετικότητα οι κάτοικοι αυτών των κρατηδίων. Και δυστυχώς υπάρχουν λίγοι, λίγες οργανώσεις ε, νέων στις οποίες να συνέρχονται παιδιά προσφύγων και μετανάστες ε, ώστε να μπορούν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να εκφράσουν τα, το τι τους ενδιαφέρει. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να εμπλακούμε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι δείχνοντας μεγαλύτερη ευρύτερη κατανόηση, ιδιαίτερα στη διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου αυτών των παιδιών και νέων, ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτές τις ομάδες στόχους. Όμως η ένταξη μπορεί να επιτύχει μόνο όταν ανοίξουμε τα θεσμικά μας όργανα και ε, εργαλεία όσον αφορά την πολιτιστική πολυμορφία. Έχουμε την έννοια του ε, πολυπολιτισμικού ανοίγματο, όπως το αποκαλούμε, εντός εισαγωγικών, που πρέπει να πολλαπλασιαστούν και να ενδυναμωθούν με κάθε τρόπο ώστε να μπορέσουν να βρουν δυνατότητες εφαρμογής και δράσης ακόμα και σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν τέτοιες εμπειρίες. Και η ένταξη σημαίνει προσωπικά να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει τις, ε, ε τις ιδεολειψίες του και τις φοβίες του, να ξεπεράσει αυτές τις φοβίες και ιδεολειψίες. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους δασκάλους, το ε, προσωπικό που έρχεται σε επαφή με αυτά τα παιδιά και αυτοί θα πρέπει να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκαταλήψεις τους και την ιδεολειψία τους ο άτυπος τομέας εκπαίδευσης, στον τομέα της πολιτικής και πολιτιστικής ε, εκπαίδευσης, στα συμβούλια αυτά των νέων πρέπει για τους νέους, από τους νέους να διαμορφώνονται. Θα πρέπει σε όλους τους ε, τομείς ε, να δημιουργηθούν οι, δομείς, δομές, να δημιουργηθούν οι συναντήσεις των νέων και να δημιουργηθούν διαδικασίες ζήμωσης και αλληλεπίδρασης που θα είναι σημαντικές για την ένταξη. Η συζήτηση για τη συμμετοχή των νέων σε όλα τα επίπεδα λήψης απόφασης που, που αφορούν τους νέους από πλευράς των αστικών κέντρων μέχρι και στο επίπεδο των κοινοβουλίων νέων συνεισφέρει για να ευαισθητοποιηθούν πολύ περισσότερο τα παιδιά αυτά και οι νέοι ε, για τη συμμετοχή τους και ενδυναμώνεται η αναγνώριση της νεότητας ως μιας φάσης στην οποία οι άνθρωποι θα πρέπει να αποκτήσουν τη δική τους φωνή και να ανακαλύψουν το ποιοι είναι και το ίδιο πρέπει να γίνει και στις ευρωπαϊκές στρατηγικές. Οι νέοι πρόσφυγες στη Γερμανία και άλλες, ε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτές τις δράσεις. Είναι σημαντικό η αξία, η πρόσθετη αξία των νέων στο εθνικό επίπεδο να μπορέσει να υλοποιηθεί. Στις περισσότερες χώρες προέλευσης ε, από τις οποίες προέρχονται τα παιδιά αυτά έχουν λιγότερα δικαιώματα. Ποιο ρόλο λοιπόν μπορούν να διαδραματίσουν οι κοινωνικά εμπλεκόμενοι ώστε να υπάρξει ανεξαρτησία, ανεξαρτοποίηση αυτών των νέων και ποιος είναι ο ρόλος των άτυπων ε, δυνατοτήτων θα πρέπει να εξηγηθεί στα παιδιά αυτά για να μπορέσουν να δράσουν με τον πιο σωστό τρόπο. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έλπιζα να είχαμε ως ε, ε, βοήθεια, μια ενίσχυση της κοινωνικής αυτής αστικής δράσης ιδιαίτερα όσον αφορά τη δουλειά που κάνουμε με παιδιά και νέους. Ενισχυμένη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα μέλη όσον αφορά την πολιτισμική, διαπολιτισμική εργασία στα κέντρα νέων και συμβούλια νέων, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε συναντήσεις, θα θέλαμε να μειωθεί η γραφειοκρατική επιβάρυνση που συνεπάγονται προγράμματα όπως το Erasmus Sin, Erasmus Plus, όπως οι για την Ευρώπη, οι ε, οργανώσει ε, που, των νέων για την ε, ε, συλλογή, για, την, για τις διαφορετικές εμπειρίες που μπορούν να δοθούν μέσω αυτού του τρόπου. Η αντιμετώπιση μιας, η προώθηση μιας εικόνας δημοκρατικής και αλληλέγγυας Ευρώπης. Η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον άτυπο αυτό τομέα εκπαίδευσης και παιδείας ώστε να γίνει αποδεκτός και να μπορεί να υποστηρίζεται. Και θα θέλαμε να έχουμε το πρότυπο μιας δημοκρατικής πολιτικής και αλληλέγγυας Ευρώπης ως βάσης της αποτελεσματικής ένταξης των ανθρώπων αυτών σε αυτήν. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε το τι θέλει η νέα γενιά και αυτό που μας είπε το Συμβούλιο Νέων είναι πολύ ε, σημαντικό και για την άτυπη εκπαίδευση και παιδεία και για ε, τις διαφορετικές ε, δυνατότητες οι οποίοι προσφέρονται. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στον, στην δόκτωρα Πεσότση για τις καριέρες των νέων μεταναστών, τις ευκαιρίες κτλ. Θα ήθελα παρακαλώ να παραμείνεις πιστή στο χρόνο γιατί Εκεί έχουμε πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Πολιτισμού και την Πρόεδρο για αυτή την ε, πρόσκληση που μου επέτρεψε να παρουσιάσω κάποιες ιδέες ε, για το θέμα της ανθρωπιστικής ε, για, το θέμα αυτό της καριέρας που είναι δυνατή παρόλο που μπροστά στην ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα θέματα δεν μοιάζουν σημαντικά. Ένα από τα πιο βασικά που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι τι συμβαίνει με την ενσωμάτωση με την ενσωμάτωση στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, εθνικές κοινωνίες γενικότερα ε, προκύπτει το θέμα του τι ακριβώς σημαίνει η θαγένεια ευρωπαϊκή και τι σημαίνει αυτό για την όμορφη ζωή την οποία ζούμε σήμερα, ίσως και αύριο. Στο ίδιο πλαίσιο ήθελα να εντάξω την προσπάθεια ανάκτησης της μνήμης, διότι εάν ξαναδούμε αυτό που έχει πει και έχει πράξει η Ευρώπη ως τώρα ως προς την ένταξη των μεταναστών, ιδίως των νέων γενεών, βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια δυνατότητα με κληρονομιά ολόκληρη, κληροδότημα μελετών, εκθέσεων, ε, μαρτυριών και του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει και μια διαφορετική πραγματικότητα ως προς τη μετανάστευση στα διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Στη μετάλλη λόγου χάρη, πρόσφατα ε, είναι πιο έντονο το φαινόμενο της μετανάστευσης, ενώ στη δεκαετία του 90 το πρόβλημα ήταν κυρίως το θέμα της ε, μετανάστευσης από την Ιταλία. Εδώ λοιπόν, ε, όπου υπάρχει και μία ιδιαιτερότητα, πολλές φορές υπάρχει και μία σύγκληση των προβληματισμών που προκύπτουν. Έτσι λοιπόν, στο κέντρο όλης αυτής της συζήτησης, η ένταξη, η συμμετοχή, ποια πρέπει να είναι η ένταξη των νέων, ποιες οι δυνατότητες ένταξης, για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όλα αυτά είναι σημαντικά θέματα. Θα άξιζε λοιπόν ακριβώς με αυτή την ευκαιρία που έχουμε εδώ να συζητήσουμε να προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε και την ιστορική μνήμη της Ευρώπης ε, υπό αυτή την προοπτική ακριβώς γιατί θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι πολλά πράγματα που τα εκφωνώ τώρα δεν είναι καινούρια έχουν ήδη συζητηθεί στην Ευρώπη λόγω χάρη με τη συζήτηση περί ηθαγένειας και την ένταξη στα σχολεία ή τον διαπολιτιστικό διάλογο. Το 2008 γιορτάστηκε το ε, ε, Ευρωπαϊκό Έτος του Διαπολιτισμικού Διαλόγου και από τότε έχουμε πολύ κέρια έγγραφα και κείμενα στη διαθέσή μας. Πέραν όμως της ιστορικής μνήμης ήθελα να φωτίσω και το όλο τοπίο αυτών των συλλογιστικών, δηλαδή το τι θα κάνουμε τις γενιές των νέων μεταναστών, τα παιδάκια που βλέπουμε και στα, στις βάρκες, στα σκάφη, ε, στη θάλασσα, στα χέρια, στην αγκαλιά των μανάδων τους, να βρίσκονται σε διέλευση να φτάνουν στην Ευρώπη. Οι γενιές αυτών των νέων ξένων μοιάζουν πολύ με τις δικές μας τις γενιές, τις γενιές των ντόπιων. Μοιάζουν διότι ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, ψηφιοποίησης, πολυπολιτισμικότητας. Όλοι αυτοί είναι ε, όσοι είναι ηθαγενείς μιας χώρας, έχουν την ηθαγένεια μιας χώρας με τον, με τον ψηφιακό διάβλο μπορεί να ανήκουν πραγματικά και σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή μπορούν να έρχονται από μια άλλη θρησκεία, γλώσσα, χώρα, αλλά η παρουσία τους μπορεί να διευθετηθεί. Αυτός είναι ένας ε, ενεργός ρόλος που μπορεί να αναλάβουν και τα σχολεία. Όμως δεν μπορούμε και να ξεχνάμε τις διαφορές που υπάρχουν. Υπάρχουν σε κάθε περίπτωση μεταξύ των νέων γενεών εφόσον πρόκειται για νέους μετανάστες ή έχουν, ε, είναι μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, όπως στη Γαλλία. Έχουν δηλαδή οικογένεια μετανάστε, που εντάσσεται στο φαινόμενο της μετανάστευσης. Εκεί διαφέρουν οι συνθήκες διαβίωσης ή και οι επιθυμίες για τη ζωή, τα σχέδιά τους για τη ζωή λόγω της ε, Πρέπει αυτές οι διαφορές λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη. Εδώ θα ήθελα να κάνω μια ουσιαστική παρατήρηση, διτή μάλιστα. Μια επιλογή που ξεκινά από μια σφαιρική προσέγγιση, όπως είπε και η κυρία Κέντζε, για τη μετανάστευση συνολικά, αλλά και για το πώς οι νέες γενιές νέων μπορεί να αντιμετωπιστούν. Σφαιρικό θα πει περισσότεροι φορείς που μπορούν να συμμετέχουν, οικογένεια, σχολείο, αλληλένδετοι μεταξύ τους, όπως έδειξαν και οι προηγούμενες εκθέσεις, ιδίως η παρουσίαση του κ. Πιατσαντίνη. Επίσης και μια δυναμική προσέγγιση, μια προσέγγιση που δεν θεωρεί τη μετανάστευση, το μετανάστη ως μια κατάσταση ιδιαίτερη, μια κατηγοριοποίηση, αλλά μια ενεξελίξη διαδικασία. Μια ενεξελίξη διαδικασία που οι νέοι άλλο ε, θα είτε έχουν γεννηθεί αλλού είτε εδώ από μετανάστες γονείς είναι σε κάθε περίπτωση, ε, μπορούν να θεωρηθούν ενεργά πρόσωπα στην όλη διαδικασία. Και εδώ ε, πρέπει να επικεντρωθούμε στη δυνατότητα των προσώπων αυτών και να λάβουν αποφάσεις και να δράσουν στο πλαίσιο συγκεκριμένων δομών πολιτιστικών και κοινωνικών. Έπειτα έχουμε κατά νου τους νέους που βρίσκονται σε φάση μεταβατική. Νέοι οι οποίοι έχουν οικογένεια ή ανήκουν ε, σε οικογένεια, σε έναν περίγυρο κοινωνικό, ένα κοινωνικό περιβάλλον μέσω της σχολικής όμως διαδικασίας μπορούν να οδεύσουν προς ένα διαφορετικό μέλλον και την εργασία. Αυτό είναι συνήθως το κλασικό προφίλ. Ένα προφίλ που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και για τους Ιταλούς, τους ξένους, τους Ευρωπαίους με τον ίδιο τρόπο. Θα πρέπει λοιπόν να ε, ληφθεί υπόψη συνολικά, αλλά για τους νέους μετανάστες όλος ιδιαίτερος και να σκεφτούμε τη δυνατότητα να ε, απαλλαγούμε από αυτό αυτές διαφορές στο βιογραφικό διακοπές ή δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουν συστηματικά οι νέοι όπως πρόσφατα έδειξε μια μελέτη του Ανδρέας Βάιτερ που συγκρίνει διαφορετικές καταστάσεις μεταξύ τους από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης. Θεωρώντας, ε, μάλλον βλέποντας το τι γίνεται στην οικογένεια μεταναστών βλέπουμε επίσης να υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία καταστάσεων διαφοροποιημένη σύνθεση οικογενειών, οικογένειες μόνο γονεϊκές με ιδιαίτερη προσοχή στους εσωτερικούς δεσμούς της οικογένειας, αλλά και με ιδιαίτερη σύνδεση με αυτά που έμειναν πίσω στη χώρα προέλευσης. Μεγάλη επένδυση στις οικογενειακές σχέσεις και στο μέλλον των παιδιών σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες αλλά και διαφορές μεταξύ ντόπιων και ξένων οικογενειών, οικογενειών μεταναστών. Η οικογένεια Λαδαπών συνήθως έχει πολλά προβλήματα παρόμοια με αυτά των δικών μας των ευρωπαϊκών κοινωνιών όμως η πορεία της μετανάστευσης έχει και πολλές επιπτώσεις ιδιαίτερως στα παιδιά. Από τις έρευνες ε, που και εγώ ίδια διεξήγαγα φάνηκε πως Είναι ελλειπής η επικοινωνία μεταξύ των ντόπιων οικογενειών και των ξένων. Σε γενικές γραμμές τα βλέμματα διασταυρώνονται, αλλά περισσότερο οι πορείες παραμένουν παράλληλες και δεν συναντώνται. Όπως είπε και ο κύριος Πιατσεντίνη με τα δεδομένα που έχει συγκεντρώσει, το προηγούμενο, το ιστορικό των νέων αυτών δεν είναι αμεληταίο. Είναι η κορυφή ενός παγόβουνου και είναι πολύ καλά κρυμμένο το υπόλοιπο παγόβουνα και όπως μας είπε και ο ΑΣΕ από το 2012 σε σχετική έκθεση. Αυτό λοιπόν δυσκολεύει πολύ τα πράγματα για τις προσπάθειές μας και εδώ το σχολείο πραγματικά μπορεί να αποτελέσει μια λύση. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2012 πολύ, πολύ σωστά ε, προέβαλε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ε, για τους μαθητές που έρχονται από το χώρο της μετανάστευσης ή έχουν ε, παρελθόν μεταναστευτικό. Το σχολείο λοιπόν μπορεί να αποτελέσει λύση, ε, είναι ένας πόρος και αυτό το δείχνουν και έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί στην Ιταλία. Ιδίως τα τελευταία 20 χρόνια για τη μετανάστευση των άλλων δαπών νέων και τη σχέση τους με το σχολείο. Οι ξένοι μαθητές ε, πολύ πρόημα ε, κατευθύνονται σε επαγγελματική κατάρτιση, όπως ονομάζεται σε εμάς στην Ιταλία, γενικότερα σε εκπαιδευτικά προφίλ χαμηλών των προσόντων. Επίση υπάρχουν πολλέ περιπτώσει σχολική αποτυχία ή σχολική καθυστέρηση. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και θετικέ σχέσει, θετικέ σχέσει με του δασκάλου και του διδάσκοντε και πολλέ φορέ σπανιότερα είναι η πρώτη τη τάξη. Μια πολύ σύντομη παρένθεση για δύο αποτελέσματα πραγματικά όμορφα στην έρευνά μα. Μια έρευνα που διεξήχθη για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τη δεύτερη βαθμίδα, η οποία εξέτασε το τι γίνεται με τους μαθητές στα γυμνάσια και τα λύκεια, στην επαγγελματική κατάρτιση και προέκυψαν τρεις βασικές κατηγορίες αυτών των χαμηλών προσόντων. Ε, η δυνατότητα της ε, αφομοίωσης, ε, της ρεαλιστικής αφομοίωσης, διερεύνησης δηλαδή και εκμάθησης. Εάν δείτε τι έχω γράψει στη διαφάνεια κάτω από το κάθε προφίλ, βλέπετε πόσο σημαντική είναι η κοινωνικονομική προέλευση, αλλά και τα κίνητρα που έχει αρχικά στον προσανατολισμό του μαθητής, ο οποίος... Ε, δεν στρέφεται τόσο πολύ στην παιδεία, αλλά περισσότερο στην εργασία. Ε, υπάρχει λοιπόν το χαμηλό αυτό προφίλ όπως λέγεται, χαμηλών προσόντων, ε, χαμηλή επένδυση, επίπεδο επενδύσεων για να ξεφύγει από την κατάστασή του. Μια δεύτερη έρευνα, πιο πρόσφατη, ε, απέναντί μας έδειξε ότι πρέπει να μετρήσουμε σωστότερα τη μετανάστευση, στα σχολεία. Και υπάρχει ένα πολύ προφανές, ένα μάλλον πολύ ε, σημαντικό αποτέλεσμα όπου υπάρχει μια κατηγορία με ελάχιστη επιτυχία και ελάχιστη ένταξη στην τάξη, αλλά και το ακριβώς αντίθετο. Εν στο μέσο υπάρχει και η μερική ένταξη. Το 35% του δείγματος των πάνω από 30.000 μαθητών που, 30.000 μαθητών που συμμετείχαν, εκεί οι Ιταλοί και ξένοι λένε ότι είναι καλά στο σχολείο παρόλο που δεν τα πάνε καλά στα μαθήματα. Είναι λοιπόν ε, άνετα γιατί είναι ε, καλά μαζί στη συνύπαρξή τους ως ομάδα συνομιλίκων, ως ε, ομότιμοι. Οδεύω προς το, την ολοκλήρωση της ομιλίας μου διότι αυτά είναι απλώς μερικές σκέψεις. Μας λένε πως η πρώτη και η δεύτερη γενιά έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Πολύ γρήγορα να θίξω και το τελικό ζήτημα που με ενδιέφερε, η ένταξη. Η ένταξη δεν μπορεί να ειδωθεί ως ένα μοντέλο ενιαίο, ένα ε, μοντέλο αφομοίωσης ή νέο αφομοίωσης ή πολυπολιτισμικό ε, με ε, πολύ πολιτισμική προσέγγιση. Αλλά θα πρέπει να την ξανασχεδιάσουμε με μια ρεαλιστικότατη εξέταση της πραγματικότητας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Με νέους δρόμους που θα πρέπει να προσανατολίζονται στον διάλογο και την πράξη όπως ε, προκύπτει στην κοινωνία, στην καθημερινή ζωή. Ο χώρος της καθημερινότητας, του σχολείου, της οικογένειας, της γειτονιάς είναι αυτά που θα να μας κατευθύνουν. Όχι λοιπόν πλέον ένα μοντέλο ένταξης ε, που καλά σχεδιάζεται στη θεωρία και επιβάλλεται ε, στη συνέχεια, αλλά ένα διαλογικό μοντέλο ένταξης το οποίο συνδιαρθρώνεται, συνσχεδιάζεται μέρα τη μέρα στους πολλαπλούς χώρους όπου ε, προκύπτει η εμπειρία και ο καθημερινός βίος. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε πολυπολιτισμικό της καθημερι... πολυπολιτισμό της καθημερινότητας. Μιλάμε για πολλές δυναμικές σχέσεις που προκύπτουν από την τριβή και την συνύπαρξη με ιδιαιτερότητες που εκφράζονται επιμέρους σε ατομικό επίπεδο αλλά μετά σε μεγαλύτερο επίπεδο σε συγκεκριμένες περιοχές, χώρους κοινωνικούς ε, και σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα. Θα ήθελα να κλείσω με αυτές τις παρατηρήσεις. Είναι μια κοινωνική πρακτική η ένταξη, γιατί μόνο έτσι δημιουργείται η θαγένεια των πολιτών, το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινωνία και σε ένα πολιτισμό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μπεζότση για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ομιλία και για την παρουσίαση των ερευνών και των συμπερασμάτων προς ένα μοντέλο που να είναι διαπολιτισμικό, πολυπολιτισμικό και να συνσχεδιαστεί από όλους τους ε, συμμετέχοντες και ενδιαφέροντες. Θα μπορούσε να συμβάλλει τα μάλα στις εργασίες μας. Να δώσω το λόγο σε όσους ε, τον έχουν ζητήσει. Παρακαλώ μεταξύ σας, μάλλον όχι, ε, εσείς στο πάνελ, εάν μπορείτε να μοιραστείτε το χρόνο που σας έχει προβλεφθεί, αλλά όσο μπορείτε πιο σύντομα μεταξύ σας για την τέχνη και τις δυνατότητες να εξυπηρετήσει την ένταξη. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, η κυρία Γκαριάτσο, δεν μπορούμε να καλούμε εδώ ανθρώπους που έχουν τέτοια εμπειρία, χωρίς να τους δίνουμε το λόγο. Η κυρία Ουαμάρη που είναι Βελγίδα επίσης και είναι προέλευσης ε, από το Μαρόκο, Βερβέρα, θα λάβει το λόγο στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ακουστεί και η δική μας μικρή φωνή, η φωνή των καλλιτεχνών που συχνά βρίσκονται μάλλον ε, στην περιφέρεια των συζητήσεων τέτοιου είδους. Εμείς λοιπόν μέσω των project του Ιδρύματος Γεχούντι Μενουχίν που έχουν παρουσιαστεί εδώ και πολύ καιρό εδώ όταν ήταν ακόμα και στην πρόεδρος της Επιτροπής ε, πολιτισμού στις αρχές της δεκαετίας του, 90 είχε έρθει ο ίδιος ο Γεχούντι Μενουχίν να μιλήσει για το δικό του ίδρωμα που τότε έκανε ένα πραγματικά καινοτόμο ε, διάλογο γιατί κανείς δεν μιλούσε τότε για τις πολιτιστικές μειονότητες Ευρώπης και ο ίδιος ήθελε να δημιουργήσει μια συνέλευση των πολιτιστικών μειονοτήτων και μειονοτικών πολιτισμών στην Ευρώπη εδώ στο Κοινοβούλιο για να μπορούν όλοι να εκφράσουν τον πλούτο τους. Τότε αυτό έμοιαζε σαν αδύνατο ε, άπιαστο όνειρο, αλλά τελικά καταφέραμε να δημιουργήσουμε αυτό το βήμα. Δημιουργήθηκε το 1991 στις Βρυξέλλες το Ίδρυμα αυτό με στόχο να δώσει φωνή σε αυτούς που δεν την έχουν μέσω projects ξεκινώντας από τα παιδιά. Οι ιδέες λοιπόν του Γιαχόντι Μενοχήν ε, που ε, επηρεάστηκε από το Ζόλταν Κονταΐδ ήταν να έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση από την πιο νεαρή ηλικία ε, στο δυναμικό τους έτσι ώστε να μπορούν με φυσικό τρόπο να εκφραστούν μέσω των συναισθημάτων τους. Ήταν πεπισμένος πως πριν μάθει ένα παιδί μαθηματικά, επιστήμες και τις πιο δύσκολες, ε, τα πιο δύσκολα μαθήματα στο σχολείο θα μπορούσε ήδη να χορεύει ε, για να αισθάνεται καλά με το σώμα του, με, τις, ε, με τα συναισθήματά του, με τα όσα τα απασχολούν και μετά να ασχοληθεί με τις ε, πιο καθαρά διανοητικές δραστηριότητες. Δημιουργήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα MUSE που είναι η μουσική και όλες οι τέχνες που διδάσκονται στο σχολείο στην Ευρώπη και ξεκινήσαμε εκεί. Γιατί είμαστε σε 13 κράτη παρόντες στην Ευρώπη με 800 καλλιτέχνες που ε, τακτικά ε, δραστηριοποιούνται στα δημοτικά. Το 10% των σχολικών ορών αφιερώνονται σε αυτό. Είναι ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο και οι καλλιτέχνες συνεργάζονται με του ε, διδασκάλους κάθε εβδομάδα τουλάχιστον για τρία χρόνια έτσι ώστε να προσφέρουν αυτά τα οποία έχουν ζήσει ω καλλιτέχνες και να δημιουργήσουν μαζί με το δάσκαλο μία καινοτόμο σχέση που θα ευνοήσει τα παιδιά. Αυτό πρόσφερε πάρα πολύ μεγάλο πλούτο και η Πατρίς Βίτσερς που είναι μία από τις μεγάλες καλλιτέχνες που έχουμε στο project αυτό θα σε εξηγήσει πώς γίνεται. Θα της δώσω το λόγο σε λίγο. Θέλω μόνο να αναφερθώ ε, στα όσα έλεγε ο Γεχούντι ε, Μενουχίν που ισχύει και για σήμερα. Ζούμε μία εποχή όπου είναι απαραίτητο να αλλάζουμε για να επιβιώνουμε. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τις ε, αντιμαχίες και να ανοίξουμε στην αλληλεγγύη, στην αμοιβαιότητα, στη συμπληρωματικότητα. Μέσω λοιπόν project σαν και αυτά τα οποία έχουμε τα καλλιτεχνικά project στα δημοτικά σχολεία θα δημιουργήσουμε την αμοιβαιότητα, την αλληλεγγύη γιατί κάθε παιδί πρέπει να ακουστεί και αυτό ισχύει και για τα παιδιά εδώ και για τα παιδιά αλλού. Όλα τα παιδιά έχουν μια εσωτερική φωνή που πρέπει να εκφραστεί. Και αν δεν δοθεί χώρος για να εκφράσουν αυτό, ε, τα παιδιά θα πληγωθούν και σιγά σιγά αυτό θα μετατραπεί σε βία, όπως έχει γίνει σε πολλά από τα γκέτο σε μεγάλες πόλεις σήμερα. Θα πρέπει στα παιδιά να δοθεί ευκαιρία από την πιο νεαρή ηλικία να εκφράζονται, να βρουν τη φωνή του. Είναι μια παιδαγωγική η οποία μέσω των τεχνών δίνει σε όλα τα παιδιά από όλους τους πολιτισμούς ε, μία διάβλο έκφρασης, ένα διάβλο έκφρασης, με συγχωρείτε, έτσι ώστε να εκφράζονται ε, και όχι απλώς να μαζεύουν αφηρημένες έννοιες οι οποίες ε, ίσως τελικά δεν θα χρησιμεύσουν στη ζωή τους για σήμερα. Σας έδειξα τα περισσότερα πόσα είχα στο PowerPoint, νομίζω έκανα μια γρήγορη σύνοψη, απλώς να σας δείξω και το πού βρισκόμαστε με το πρόγραμμα Μούσα σήμερα. Να οι χώρες, 12 χώρες και το Ισραήλ και στα διάφορα σχολεία έχουμε συνολικά πλησιάσει 40.000 παιδιά με διαφορετικούς τρόπους. Σε κάποια κράτη τα project ακολουθούν άλλη εξέλιξη, αλλά βλέπετε εδώ πώς είναι οι καλλιτέχνες που συνεργάζονται μαζί μας συχνά σε συνεργασία με τους δασκάλους. Και τώρα το λόγο έχει μια καλλιτέχνηση η οποία θα σας εξηγήσει ακριβώς πώς γίνεται σε καθημερινό επίπεδο με τα παιδιά σε μια αίθουσα σχολική στο Βέλγιο. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. I'm a second generation. Είμαι δεύτερη γενιά στο Βέλγιο. Έφυγαν, διώχθηκαν από την Ινδονησία οι γονείς μου και στο σπίτι με αυτό με ανανούριζαν. Ελπίζω να μην σας κοίμησα. Και με τέτοιους, ε, με, με καραγκιόζι παίζαμε στους τοίχους. Και όταν ερχόντουσαν Ολλανδοί να μας επισκεφτούν, ε, τα κρύβαμε, δεν μιλούσαμε τη γλώσσα μας. Οπότε αυτή ήταν η πολιτική των γονιών μου έτσι ώστε εμείς να αφομοιωθούμε, έτσι λεγόταν τότε, και λυπάμαι τόσο πολύ. Και σαν καλλιτέχνη υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως εγώ θέλω να δώσω στα παιδιά τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν διαφορετικά στα σχολεία. Θα πρέπει να καλωσορίζουμε το γεγονός πως τα παιδιά μπορούν να τραγουδήσουν σε διαφορετικές γλώσσες, να μιλήσουν διαφορετικές γλώσσες, να φέρουν τον πολιτισμό τους μαζί, γιατί αυτό είναι πλούτος και ήμουν τόσο χαρούμενη όταν βρήκα το δίκτυο Μούζε που μου επέτρεψε να εξελίξω κάτι τέτοιο ως καλλιτέχνης στην πρώτη αυτή διαφάνεια βλέπετε το δίκτυο Μούζε το οποίο οργανώνει πολλές συναντήσεις μεταξύ καλλιτεχνών διεθνών καλλιτεχνών και πρέπει να σας πω ότι μου εξήγησαν διάφορες μεθόδους, τις οποίες εγώ στην τάξη μέσα εφαρμόζω. Για παράδειγμα, στη μεσαία φωτογραφία βλέπετε ένα τραπέζι ζωγραφισμένο με πολλά διαφορετικά εδέσματα και το έφερα στο Βέλγιο και είπα, ας αφήσουμε όλα αυτά τα παιδιά, παρόλο που έχουμε, για παράδειγμα, 10 διαφορετικά ε, πολιτικά υπόβαθρα σε μια τάση με 20-24 παιδιά, γιατί να μην τους επιτρέψουμε να φέρουν τις συνταγές τους από το σπίτι και τα ε, όσα χρησιμοποιούν στη μαγειρική στο σπίτι τους ε, και να μαγειρέψουμε, να ζωγραφίσουμε ε, με τα μπαχαρικά γιατί βέβαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως χρωστικές ε, και να φέρουμε μια νέα δυναμική στο σχολείο ένα τρόπο νέο εκμάθησης όχι μόνο για τα παιδιά μεταναστών αλλά και για τα υπόλοιπα γνωρίζουμε και ε, μαθαίνουμε ένας από τον άλλο είναι διαφορετική μέθοδη άτυπης εκπαίδευσης σε ένα άτυπο περιβάλλον εκπαιδευτικό και μαθαίνουν μαζί και οι δάσκαλοι. Γιατί οι δάσκαλοι είναι η βασική μας εταίροι για να είναι επιτυχημένο αυτό το project και μαζί με αυτούς το περνάμε και στο πιο επίσημο επίπεδο γιατί έχει να κάνει με τα μαθηματικά, με τη γλώσσα, με πολλά. Είναι η τέχνη, είναι η κοινωνική δεξιότητα, είναι η συναισθηματική ε, γνώση. Είναι μια ολιστική προσέγγιση λοιπόν. Μία ακόμα διαφάνεια με κάτι που κάνω αρκετά συχνά στην τάξη ως καλλιτέχνης είναι να αφήσω τα παιδιά να φέρουν αντικείμενα από το σπίτι. Για σας τι είναι αντικείμενο από το δικό σας πολιτισμό. Μπορεί να είναι πάρα πολλά. Μπορεί να είναι ρούχα. Μπορεί να είναι ε, κεραμικά, μπορεί να είναι κοσμήματα. Τα φέρνουν στο σχολείο και μας τα παρουσιάζουν. Και για το τι σημαίνουν καμιά φορά είναι κομμάτι του πολιτισμού τους και δεν γνωρίζουν τι εκπροσωπούν και ψάχνουμε μαζί στο διαδίκτυο να βρούμε τι σημαίνει και αυτό είναι και διασκεδαστικό γιατί όλα πια μπορείς να τα ψάξεις στο ίντερνετ. Και στο project αυτά τους αφήνουν να ζωγραφίσουν τα αντικείμενά τους και έχουμε ε, φράχτες που είναι 20 μέτρα και ήρθαν οι γονείς και τα είδαν ζωγραφισμένα και είπαν πω πω αυτό το αναγνωρίζω και εκείνο το αναγνωρίζω και είναι σαν να γυρίζω σπίτι μου παρόλο που είμαι στο σχολείο είναι σημαντικό αυτό λοιπόν. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι γονείς έτσι ώστε να γίνεται και ένας διάλογος μαζί τους. Εγώ οργανώνω ατελιέ, εργαστήρια με τα παιδιά, ένα χρόνο τουλάχιστον με όλα τα παιδιά σε μια τάξη. Και οργανώνω επίσης τώρα και ατελιέ μόνο με τους γονείς και μετά με γονείς και παιδιά μαζί. Το project μουζέ είναι κυρίως για τα δημοτικά, αλλά όλο και περισσότερο περνάμε και σε γυμνάσια με τους νέους και τις νέες που σε λίγο θα είναι οι ενήλικες του μέλλοντος και θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα είναι περιορισμένος ο χρόνος η μουζέ επίσης ε, πηγαίνει σε ε, προσφυγικούς καταβλισμούς με ανήλικα που ε, το έσκασαν μόνα τους από, τον, ε, από τη χώρα τους και πολλές φορές τους ρωτάμε πάνω στο χάρτη δείξε μου πώς πήγες από το Αφγανιστάν στο Βέλγιο και σου δείχνουν στο χάρτη και δεν έχουν να την πιο σύντομη οδό. Είναι πραγματικά, κάνει κύκλους με φρικτά πράγματα. Έχουν εκπορνευθεί. Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ε, πώς οι έφηβοι αυτοί έφτασαν στο Βέλγιο με τέτοιους τρόπους. Αυτό το αφήνω τώρα. Ως καλλιτέχνης ή ως καλλιτέχνες, γιατί εδώ εκπρόσωπω τους πολλούς καλλιτέχνες στο δικό μας project, το Μούζε, επιτόπου αλλάζει συνέχεια η κατάσταση και χρειάζεται να συλλέξουμε κάπου τις βέλτιστες πρακτικές για να τις μοιραστούμε με τους υπόλοιπους και είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι σήμερα εδώ και σας περιγράφω τι κάνουμε στο δίκτυο για χούντι Μενουχίν τη μεθοδολογία που ακολουθούμε και ελπίζω πως θα μπορέσουμε να τη μοιραστούμε όλο και περισσότερο με άλλες οργανώσεις. Έχω 15 χρόνια, 16 μάλλον, που εργάζομαι στο πρόγραμμα αυτό, ποτέ δεν έχω βαρεθεί και είμαι ακόμα φίλη με ένα από τα παιδιά που είχα σε μια από τις τάξεις μου πριν από 10-12 χρόνια και θέλω να της δώσω το λόγο. Που είναι πια μια όμορφη νέα κοπέλα. Φάρα Yes, okay. Uh, thank you, Patrice. Ευχαριστώ πολύ Πατρίς που με κάλεσες. Είμαι 23, λέγομαι Φάρα Λομάνη, οι γονείς μου είναι από το Μαρόκο, οπότε φαντάζομαι αυτό με κάνει Μαροκινή. Εμείς κάναμε μιούζες στο δημοτικό και το θυμάμαι ότι όταν ήμασταν δημιουργικοί η μόνη γλώσσα που μιλούσαμε ήταν η γλώσσα της δημιουργικότητας, της εκφραστικότητας, της δημιουργίας. Θυμάμαι να διασκεδάζουμε, να μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και να σεβόμαστε τις διαφορές αλλήλων και τις παραδόσεις αλλήλων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Οπότε έχουμε δύο γενιές γυναικών με διαφορετική ιστορία ένταξης και βρήκαν τη φωνή τους για να εκφραστούν, πράγμα που συνδυάζεται και με όσα μας είπε η δασκάλα μας προηγουμένως για το σχολείο. Το σχολείο όμως δεν είναι απομονωμένο, εάν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες ένταξης, συνοδείας και ε, παρακολούθησης. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ομιλίες. Έχουμε κάνει πολύ σοβαρή δουλειά σήμερα με όλες αυτές τις πληροφορίες και μας δώσατε πάρα πολλές πολύτιμες προτάσεις και συστάσεις πολύτιμες για τη δουλειά μας. Να δώσω τώρα το λόγο να δώσω τώρα το λόγο στην δοκτόρα Καριάτσο για την οποία η μετανάστευση είναι μια προτεραιότητα, ε, μάλλον ο πολιτισμός είναι μια προτεραιότητα για την πολιτική μετανάστευση, καθώς είδαμε πρόσφατα και αύξηση των κονδυλίων για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Ζητήσαμε να διπλασιαστεί τουλάχιστον το ποσοστό και ε, καταφέραμε να έχουμε 60 εκατομμύρια για φέτος. Υπήρξε μια σχετική έκκληση στο Erasmus Plus και στη Δημιουργική Ευρώπη προς τις ενώσεις, προς τις ομάδες για αυτό το σκέλος της πολιτιστικής και δημιουργικής ένταξης, ώστε διακρατικά να ε, επεκταθούν οι καλές πρακτικές και η αριστεία σε αυτό το τομέα. Νομίζω το θέμα έχει τεθεί. Δεν μπορούμε πλέον να σκεφτούμε θα, προλαβαίν, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη εξέταση της θέματος μετανάστευσης στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια. Αλλά αυτό δεν γίνεται αν δεν τονωθεί η διάσταση της εκπαίδευσης του διαπολιτιστικού διαλόγου και της κοινωνικής ένταξης. Αρκεί να υπάρχει αλληλοσεβασμός στο πολιτιστικό επίπεδο και στις πολιτιστικές διαδικασίες και ζυμώσεις. Ευχαριστούμε για την παρουσία σα και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ που προσκαλέσατε και εμένα σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ε, εγκρόση μας εμπνέει τόσες πολλές ιδέες. Πραγματικά βλέπουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα το εκπαιδευτικό σύστημα. Πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες διέσχισαν, μάλλον έφτασαν στην Ευρώπη το 2015 και ακόμα 130.000 άνθρωποι έχουν φτάσει στην Ευρώπη διαθαλάσσης από την αρχή της φετινής χρονιάς. Και αυτό παρά τις αντικσότατες συνθήκες. Ε, το πρόβλημα λοιπόν τώρα της Ευρώπης επιβαρύνεται διότι οι περισσότεροι τους άσυλο είναι χαμηλών προσόντων ε, σε ενεργή ηλικία ή παιδιά που έχουν μείνει εκτός του σχολικού συστήματος για πολύ καιρό πριν φτάσουν εδώ. Περίπου 30% των ετούντων άσυλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015 ήταν νεότεροι από τα 18 και περίπου η μισή ήταν μεταξύ 18 και 34. Επιπλέον και παρά την έλλειψη χειροπιαστών δεδομένων, μεγάλος αριθμός ανελίκων έρθαν στην Ευρώπη ασυνόδευτοι. Στη Σουηδία, 33% των ετούντων άσυλων που έχουν καταγραφεί το 2015 είναι κατά των 18 και από αυτούς 50% είναι ασυνόδευτα ανήλικα. Είναι σαν να λέμε 35.000 μικρά. Εδώ λοιπόν η εκπαίδευση είναι το πιο ισχυρό όπλο για να δώσουμε στους μετανάστες και πρόσφυγες τα σωστά προσόντα για να πετύχουν την προσωπική τους ε, πρόοδο, να βρουν δουλειά να συμμεριστούν τις αξίες ολόκληρης της κοινωνίας και να ε, προχωρήσουν στο διαπολιτισμικό διάλογο για να μπορέσουν να περάσουν και σε ένταξη. Αυτά είναι οι βάσεις για την κοινωνική ένταξη και την ενίσχυση του ανθρωπινού κεφαλαίου μιας γυράσκουσας Ευρώπης. Εδώ λοιπόν η κατεπήγουσα εντολή μας είναι να, και καθήκον μας να εντάξουμε τους χιλιάδες πρόσφυγες στην, ε, κατεξοχήν, ε, στο κατεξοχήν εκπαιδευτικό μας σύστημα στο δυνατόν συντομότερα και οι αιτούντε άσυλο πρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα από τα πρώτα στάδια τη παιδική ηλικία, ε, στον νοικιαγωγία, στα σχολεία, στην επαγγελματική κατάρτιση, στα ανώτατα ιδρύματα και την ε, κατάρτιση των ενηλίκων για να έχουν τι απαραίτητε δεξιότητε και να αποφύγουν την περιθωριοποίηση και τη φτώχεια. Προτεραιότητα λοιπόν η ένταξη ε, θα επαφιόμαθα στην εκμάθηση γλωσσών, ακούσαμε πολλά γι' αυτό σήμερα, πόσο σημαντικό είναι. Η υποτίμηση των γνώσεων των αφιχθέντων μαθητών, οι βασικές δεξιότητες των παιδιών που είναι σε χαμηλό επίπεδο γιατί έχουν μείνει εκτός εκπαιδευτικού συστήματος πολύ καιρό όπως είπα και όπως ακούσαμε Και η διδασκαλία. Ε, η δεύτερη προτεραιότητα είναι να αποφύγουμε την αποτυχία των μεταναστών και να τους επιτρέψουμε να εκμεταλλευτούν το δυναμικό τους. Από προηγούμενα μεταναστευτικά κύματα τι διδαχτήκαμε. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες προκλήσεις. Εδώ είδαμε ότι υπάρχουν ε, σαφείς αποδεικτικά στοιχεία ότι η εκπαιδευτική επιτυχία των περισσότερων μεταναστών ε, είναι χαμηλότερη από τους συνομιλίκους της ε, συνομιλίκους τους υποδοχή. υποδοχής. Και έτσι δυσκολεύει η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και παραμένει το χάσμα δεδομένων. Ε, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι νέοι με μεταναστευτικό παρελθόν ε, κατά 70% μπορεί να οδηγηθούν σε σχολική αποτυχία και να καταλήξουν το σχολείο σε σχέση με τους ντόπιου. Και αυτό στη χώρα διαμονής μόνο και μόνο λόγω των μειονεκτημάτων στο σχολείο. Το πρόβλημα τη χαμηλή επιδόση στο σχολείο, τα βασι... χαμηλά βασικά προσόντα και την εγκατάλειψη του σχολείου σε πρώιμη ηλικία, αυτά ε, έχουν περισσότερο να κάνουν με τα κοινωνικά και οικονομικά ε, προβλήματα που είναι ε, γνωστά έτσι και αλλιώ πρώτοι η μετανάστευση η πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Εάν είναι λιγότερο μορφωμένοι από τους ντόπιου οι μετανάστε. Υπάρχουν παρόλα αυτά διαφορέ μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία, υψηλά προσόντα ε, και μεγαλύτερο πληθυσμό. Γαλλία και Ολλανδία, χαμηλότερο προσόντα μετανάστες. Ισπανία και Ιταλία. Κατά μέσο όρο δεν υπάρχουν σοβαρέ διαφορέ μεταξύ ε, εκπαιδευτικού επίπεδου ε, ξένων και ντόπιων. Ε, Πάντω, στι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε τα προηγούμενα μεταναστευτικά κείμενα έχουν οδηγήσει σε σοβαρή διάκριση και κατακαιρματισμό των προσόντων και των ε, δεξιοτήτων. Οι νέοι μετανάστε έχουν ε, επικεντρωθεί. Έχουν συγκεντρωθεί μάλλον εκτό πόλεων, σε μειονεκτούσε περιοχέ και μιλάμε για παιδιά Μαθητέ που πηγαίνουν στο σχολείο χωρί να μιλάνε τη γλώσσα τη χώρα αποδοχή. Αυτά είναι ε, γεγονότα και πρέπει να λάβουμε μέτρα για να αποφύγουμε τα λάθη λάθη που είχαμε κάνει στο παρελθόν και να αποφύγουμε να ξανασυμβούν. Εξίσου σημαντικό να αποφύγουμε την, τον κοινωνικό αποκλεισμό και να ε, καλλιεργήσουμε τον διαπολιτισμικό διάλογο με πολλές μορφές εταιρικών σχέσεων όπως ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και οι δράσεις της νεολαίας αλλά το ίδιο και η άτυπη και επίσημη εκπαίδευση. Εάν θέλουμε μια συνεκτική Ευρώπη, πρέπει ο πολιτισμό να γίνει βασική παράμετρο. Όλοι μπορούν να συμβάλλουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό, με συμμετοχή ιδρυμάτων, κοινωνικών εταίρων και κοινωνία των πολιτών. Η εργασία των νέων είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Σημαντικό στοιχείο που ε, συμβάλλει σε κοινωνίε συνεκτικέ τη συμμετοχή των ε, νέων στην κοινωνία και την αποφυγή επικίνδυνων συμπεριφορών. Σήμερα 10% του πληθυσμού της Ευρώπης έχει παρελθόν μεταναστευτικό. Αλλά οι μετανάστες της Ευρώπης επίσης συμβάλλουν ε, ιδιαίτερα στην οικονομία, τη δημιουργία ε, θέσεων απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης. Το σημερινό λοιπόν φαινόμενο, όπως είπαμε, μας είναι γνωστό από παλιά. Απλώς είναι η πρώτη φορά που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε τέτοια κλίμακα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιε ροέ προσφύγων με αριθμητική ε, διόγκωση, αλλά έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις γνώσεις μας από προηγούμενες εμπειρίες και να βελτιώσουμε τις αποκρίσεις μας, κινητοποιώντας τα σημερινά εργαλεία και προγράμματα για την καλύτερη ε, ένταξη των προσφύγων. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο, γιατί εμείς ε, και η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση ΕΑΚ, εκπαίδευση και πολιτισμός έχει αρχίσει ήδη να ενεργοποιεί τα εργαλεία που διαθέτουμε και έχουμε κάμποσα. Αναφέρατε ήδη το Erasmus Plus. Ε, ακόμη ε, την κρίση των προσφύγων και τη προκλήση της μετανάστευσης τις αντιμετωπίζουμε, της ένταξης μάλλον, τις αντιμετωπίζουμε υλοποιώντα προγράμματα που δεν άρχισαν όμως τώρα. Εάν δείτε τη βάση των δεδομένων των προγραμμάτων που έχει στηρίξει το Erasmus Plus και τα προηγούμενα προγράμματα θα βρείτε 200 παραδείγματα επιτυχημένων προγραμμάτων. Προγράμματα με αθλητισμό, αθλητικές δραστηριότητες, ε, εθελοντισμό στην, στον αθλητισμό, πολιτιστικά προγράμματα, ε, προγράμματα για την νεολαία, ε, τις διαπολιτιστικές ανταλλαγές. Η βάση των δεδομένων λοιπόν αυτή είναι δημόσια και θα σας καλούσα να ρίξετε μια ματιά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus Plus ήδη προέβλεπε το 2016 την καλλιέργεια πολιτισμικών και διαπολιτικών δραστηριοτήτων μια από τις πρώτες προτεραιότητες του προγράμματος και γι' αυτό διαθέσαμε ένα χαρτοφυλάκιο για τα προγράμματα συνεργασίας που φτάνει στα 400 εκατομμύρια ευρώ στον τομέα της εκπαίδευσης, της ε, παιδείας, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Μια από τις πρώτες προτεραιότητες για όλα τα προγράμματα που θα ασχολούνταν με αυτές τις προτεραιότητες κοινωνικής ένταξης. Επίσης έχουμε δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προγράμματα στήριξης όπου απασχολούνται μετανάστες, πρόσφυγες, ατούντες άσυλο ή την αντιμετώπιση του θέματος της κρίσης των προσφύγων γενικότερα. Επιπροσθέτως, έχουμε τώρα ένα διαγωνισμό αξίας 13 εκατομμυρίων για να ε, τόνωθούν εκατοντάδες δράσεις που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο τάξεων ε, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μια για να καλλιεργήσουμε την ένταξη των μειονεκτούντων μαθητών, ιδίως αυτούς που έχουν ένα μεταναστευτικό παρελθόν, και από την άλλη να προωθήσουμε την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και την, ε, ε, την καλλιέργεια των δημοκρατικών αξιών. Αυτό με όλα τα δημοσιονομικά εργαλεία και με τους ε, ε, εργαζομένους και το ενδιαφερόμενο προσωπικό. 100.000 άδειες δόθηκαν χρηματοδοτούμενες από τα ε, μη δαπανημένα κονδύλια των προηγούμενων ετών για την αποτίμηση των γλωσσικών γνώσεων και την διεξαγωγή γλωσσικών μαθημάτων για τους νεοφυχθέντες μετανάστες. Για μια τριετία. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη επίσης συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και θα έχουμε χρηματοδότηση για πολιτιστικές πρωτοβουλίες ώστε να υλοποιηθεί στην πράξη ο διαπολιτισμικός διάλογος και η ένταξη των ε, μεταναστών. 1,6 εκατομμύρια, μάλλον ένας διαγωνισμός αξίας 1,6 εκατομμυρίων ευρώ θα ε, προκηρυχθεί. Επίσης, η συνεργασία μεταξύ συνομιλίκων, και αυτό είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο και αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή και προβλέπουμε και δυνατότητες να δοθεί προτεραιότητα ακριβώς στον εθελοντισμό. Σε επίπεδο πολιτικής, εάν μου επιτρέψετε, πολύ σύντομα να το θίξω και αυτό, Ήδη έχουμε καταβάλει προσπάθειες για νέες δράσεις, ιδίως την εκμάθηση των ε, συνομιλίκων, την καλλιέργεια καλών πρακτικών και την ανάπτυξη καταθυντηρίων γραμμών για να στρίξουμε τα κράτη-μέλη να εντάξουν τα παιδιά στην ε, βασική εκπαίδευση. Εδώ λοιπόν η συμβολή μας είναι να διευκολύνουμε την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα με την εκμάθηση των γλώσσων και την ανάπτυξη των, των γλωσσών και την ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων και εδώ να έχουμε την ένταξη των νομίμων μεταναστών. Είπατε και εσείς κυρία Κέντζε νωρίτερα το ίδιο. Εδώ λοιπόν συμβάλλουμε στον τομέα του πολιτισμού και της παιδείας και της νεολαίας με την πρόσβαση στην εκμάθηση γλωσσών, την στήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού για να υπάρχει συμμετοχικότητα και να αποφύγουμε τη σχολική αποτυχία, αλλά και να προωθήσουμε την διαπολιτισμικότητα, τον αθλητισμό και την ε, ενεργοποίηση των νέων. Αξιοποιούμε τα εργαλεία όπως τη διδημοποίηση σχολείων, τη συνεργασία σχολικών ιδρυμάτων και την παροχή κουτιών εργαλείων για να γίνουν συγκεκριμένε συστάσει προ τα κάτι μέλη. Εν τέλει, να ολοκληρώσω με τη δήλωση των Παρισίων. Τη γνωρίζετε. Πριν από ένα χρόνο, ακριβώς πριν ένα χρόνο, η δήλωση υπεγράφει από τους Υπουργούς Παιδείας με τη συμμετοχή και του Αρμόδιου Επιτρόπου και έκανε έκκληση για την κινητοποίηση του εκπαιδευτικού τομέα σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να ε, υπάρξει μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών για τις θεμελιώδες αξίες της Ευρώπης και τις δημοκρατικές της αξίες. Είμαστε στη φάση υλοποίησης αυτής της δήλωσης. Έχει τέσσερις διαστάσεις και παραμέτρους θέλουμε να έχουν περισσότερες δεξιότητες διαπολιτισμικές, διαπολιτιστικές και ε, πολιτικές οι νέοι, το σχολικό σύστημα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα των των νέων και να προωθήσουμε το διαπολιτισμικό διάλογο και όλες τις μορφές μάθησης. Η μνήα των 30 εκατομμυρίων και του σχετικού διαγωνισμού και των 400 εκατομμυρίων του Erasmus Plus σκοπό έχουν ακριβώς να οδηγήσουν στην υλοποίηση αυτές τις δηλώσεις των Παρισιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες τελευταίες διευκρινήσεις. Ήθελα να μπορέσετε να τοποθετηθείτε όλοι στο πάνελ πρώτα, πριν ε, εκφραστούν απορίες. Και εμείς έχουμε την εξής ανησυχία. Από τη μια έχουμε πολιτικές και προγράμματα. Απ' την άλλη, Πρέπει να προσέξουμε και ελπίζω και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το καταλάβει αυτό, ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στι εκπαιδευτικέ πολιτικέ, να τι προκοδοτήσει και με τα απαραίτητα κονδύλια. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε ότι στο πρόγραμμα Εράσμου, στο πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη προβλέπονται κάποιε γραμμέ που θα αποσιωθούν σε τέτοια προγράμματα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι θα υπάρξουν και πρόσθετα κονδύλια. Όχι μόνο αυτά που ήδη προβλέπεται να εκμεταμιευθούν. Αυτά που έχουν δεσμευτεί. Διότι φιλόδοξη, το φιλόδοξο θεματολόγιο τη μετανάστευση, αυτή η νέα ανακοίνωση που περιμένουμε, η δήλωση επίση των Παρισίων, όλα αυτά πρέπει να μα κάνουν να ξανασκεφτούμε τι προτεραιότητε του προπολογισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τα σκεφτεί αυτά. Συμφωνείτε πάρα πολύ, φαντάζομαι μαζί μου. Και θα πρέπει ακόμη και στα πλαίσια των προτεραιοτήτων Γιούνκερ να φροντίσουμε να έχουμε μεγαλύτερη προσοχή και να στηρίζουμε αυτές τις πολιτικές. Ζητώ πραγματικά χίλια συγγνώμη και από εσά και από τους επικεκλημένους μας, αλλά έχω μια σημαντική τελετή στην οποία πρέπει να συμμετάσχω αμέσως τώρα. Η Αντιπρόεδρος Τρούπελ όμως θα αναλάβει την Προεδρία για να ολοκληρώσει μαζί σας και με την άλλη Αντιπρόεδρο Σοϊντρόβα και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα προεδρεύσουν λοιπόν, καθώς ξεπεράσαμε λίγο το ωράριο που προβλεπόταν. Σας ζητώ χίλια συγγνώμη, ευχαριστώ και πάλι τους προκεκλημένους και τους προκεκλημένους. Είναι πραγματικά ε, κέρια τα ζητήματα που εξετάσαμε. Εδώ δεν υπήρξε αμερόληπτη επιλογή των προσκεκλημένων, διαλέξαμε τα πιο ενδιαφέροντα βιογραφικά. Και δείχνει αυτό πόσο μεγάλη προσοχή δίνουμε στο μέλλον και τη στρατηγική εξέλιξη της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ και πάλι, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα μαζί μα και σας εύχομαι καλό βράδυ, ευχαριστώ που ήρθατε να με αντικαταστήσετε και θα φύγω τώρα. Αγαπητοί ομιλητές, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ και πάλι για τι τόσο ενδιαφέρουσε παρουσιάσει που μα κάνατε. Έχουμε τώρα χρόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Παρακαλώ για ένα λεπτό ερωτήσεις γιατί ξέρετε πως πιέζει το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Σιόντροβα έχει το λόγο πρώτη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, Λυπάμαι πολύ που έχουμε τόσο λίγο χρόνο στη διάθεσή μας για να κάνουμε ερωτήσεις και για να σχολιάσουμε, μια και πρόκειται μια ερώτηση πολύ σημαντική για μένα για την ενσωμάτιση. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως γνωρίζουμε πως ένα 38% των προσφύγων είναι παιδιά. Θα πρέπει λοιπόν να μιλάμε και για το 62% που είναι ενήλικες και οι οποίοι επίσης χρειάζονται βοήθεια για να μάθουν γλώσσες, γιατί πρέπει να μπορούν να γίνονται και αυτοί κατανοητοί. Χαίρομαι λοιπόν που μίλησαν για παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών, αλλά θα ήθελα να επανέλθω στα όσα είπε η συνάδελφος κυρία Μπάλμπεχ, γιατί είπε πως ε, είναι σημαντικοί οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι φέρουν όλο το βάρος ε, των μαθητών που χρειάζεται να ενσωματωθούν και θα πρέπει να μάθουν τα βασικά που τους χρειάζονται. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το Erasmus Plus είναι μόνο για όσους έχουν επιτυχία γιατί κάθε διευθυντής θα πρέπει να προετοιμάσει ένα project, μια αίτηση και μετά να περιμένει χωρίς τη βεβαίωση για το αν θα λάβει την χρηματοδότηση ή όχι. Η ενσωμάτωση των ε, μαθητών και η διδασκαλία των γλωσσών είναι κάτι που απαιτείται από τους καιρούς μας και δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην τύχη του. Τα σχολεία θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν πώς θα λάβουν χρηματοδότηση και αυτό ε, δεν θα πρέπει ε, να το ξεχνάμε ε, με, για το Erasmus Plus να μην κινδυνεύει και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως το Erasmus Plus δεν αποτελεί λύση για την ενσωμάτηση εκατοντάδων χιλιάδων νέων και ενηλίκων που πρέπει να μάθουν ξένες γλώσσες και πρέπει να μάθουν και τον πολιτισμό και την κουλτούρα και την κοινωνία στην οποία έφτασαν και να μάθουν πράγματα τα οποία για τους ίδιους είναι καινούργια. Αυτά λοιπόν για ε, για όλους απαιτεί χρηματοδότηση. Ευχαριστούμε πολύ για το Erasmus Plus, αλλά αποτελεί ένα πρόγραμμα συμπληρωματικό, το οποίο μπορεί να βοηθήσει αλλά δεν μπορεί να αποτελέσει τη βάση που θα χρησιμοποιούν τα σχολεία. Και θέλω για μια φορά ακόμα να ευχαριστήσω την κυρία Μπάλμπεχ που είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι δάσκαλος και χρειάζεται να τα αντιμετωπίσει. Τη θαυμάζω και θέλω ε, ε, να τη βοηθήσουμε. Νομίζω ότι ήταν μάλλον μια γενικότερη πολιτική τοποθέτηση αυτό. Τώρα, ο κύριος Μοργάνο για ένα λεπτό παρακαλώ. Πολύ σύντομα, γιατί τέτοια ώρα που πήγε δεν μπορούμε να ξαναρχίσουμε από την αρχή με μερικά ζητήματα που είναι κέρια σημασία, όπου εκεί η όλη η μελέτη θα μπορούσε να κρατήσει ώρα. τεσσερι παρατηρησει να κάνω μόνο. Νομίζω ότι πολύ σωστά η δόκτωρ Γκαλιάτσο έθεσε σωστά τι προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. στην κατεύθυνση τη ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στι άτυπε και επίσημε μορφέ εκπαίδευση λιμένος μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αν δεν δώσουμε προσοχή σε αυτό δεν θα επιλύσουμε τίποτα. Το θέμα της γλωσσικής εκμάθησης βεβαίως είναι μια πρώτη λύση. Μαζί την αφομοίωση, την αποτίμηση των γνώσεων των μαθητών που έχουν εγκαταλείψει το σχολικό σύστημα από καιρό. Υπάρχει και ένα πρόβλημα της τη του εκπαιδευτικού προσωπικού και εκτός από την ειδική κατάρτιση Υπάρχει και πραγματική υποστήριξη άλλου επίπεδου. Δεν μπορούμε τα πάντα να τα αφήνουμε στην ευθύνη του σχολείου. Επίσης για όσα μπορούν να πραγματοθούν μεταξύ συνομιλίκων, δηλαδή οι μαθητές μεταξύ τους τι μπορούν να κάνουν, αυτό μου φαίνεται ένα στοιχείο σημαντικό. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Θα Θαγένεια και και του πολίτη πάνε μαζί. Να στραφώ ε, εντάχει και στα θέματα που, που έθεσε εδώ η καθηγήτρια Μπεζότσι. Με τρεις μνήες. Πρώτον, η πρόσκληση που έγινε σήμερα βάσει των πραγματικών γεγονότων να μην σκεφτόμαστε άκαμπτα και αδιάλακτα σε ένα μοντέλο που θα μπορεί να εφαρμοστεί πανομοιότυπα παντού. Υπονοώντα τα όσα γίνονται σε επίπεδο υποδοχή και ένταξη. Αυτό μου φαίνεται καθοριστική σημασία, καθώ και οι ίδιοι έχουμε βασιστεί στην αρχή της πολυμορφίας. Δεν μπορούμε λοιπόν να σκεφτόμαστε ότι θα υπάρξει μια ενιαία λύση που μπορεί να εφαρμοστεί σε στενό σκορσέ σε όλους. Εδώ λοιπόν μου κάνει νοήματα η Πρόεδρος Κλίνο ε, πρέπει να γίνουν προσπάθειες όχι μόνο για να έχουμε ένα τέτοιο πολυ... ένα τέτοιο μοντέλο πολυμορφίας, αλλά να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη και για την υλοποίηση των ε, αρχών μας, περίπτωση την περίπτωση. Ποιος θα θέλετε να απαντήσει. Ορίστε. Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τα όσα είπατε. Νομίζω πως το Erasmus Plus όντως δεν μπορεί να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις και κάποιες από τις προκλήσεις θα πρέπει να τις απαντήσουμε εμείς. Επίσης έχουμε, έχουμε εργαλεία και στο πρόγραμμα μπορούμε να προσφέρουμε, όπως είπε και η κυρία Κώστα προηγουμένως, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών. Για το πρόγραμμα νομίζω πως αυτό το οποίο μπορεί να φέρει το Erasmus Plus είναι πρώτα απ' όλα μιλάμε για διασυνοριακή ε, συνεργασία και για τη δυνατότητα ε, ε, του να μαθαίνουμε ε, από τα όσα έχουν βιώσει όλοι. Τη στιγμή που παρουσιάζουμε τα project προσφέρουμε δυνατότητες για παράδειγμα τους δασκάλους να μάθουν από άλλους δασκάλους σε σχολεία, να συμμετέχουν σε project με άλλα σχολεία, με νέους, να συνεργάζονται με άλλους νέους και επίσης έχουμε και αυτό το νέο στοιχείο στο Erasmus Plus που είναι ε, και κάποια διακλαδικά όπου μπορούν οι σχολεία να συνεργάζονται με πανεπιστήμια ή με ενώσεις, με οργανώσεις από το χώρο του αθλητισμού. Οπότε έχουμε επίσημη και ανεπίσημη άτυπη ε, επαιδεία που μπορούν να ε, συνδυαστούν. Ένα ακόμα στοιχείο είναι το τι γίνεται σε επίπεδο πολιτικής, γιατί εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ περιορισμένες αρμοδιότητες για την παιδεία και για την εκπαίδευση. Εκεί προσφέρουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία που έχουν άλλα κράτη μέσω του peer learning, δηλαδή τις, ε, όπου τους ομολόγους τους. Έχουμε τέτοια προγράμματα που σίγουρα θα τα έχουμε για, τα συνόδευτα, για τους ανηλίκους, για τις εμπειρίες που έχουν αποκτήσει τα κράτη-μέλη από διάφορα προγράμματα και θα ανταλλαγούν αυτές οι εμπειρίες έτσι ώστε να διδαχθούμε όλοι από τους υπολείπους και η συνεργασία αυτή να φέρει ε, αποτελέσματα σε διαφορετικά επίπεδα και στο ευρωπαϊκό αλλά και στο εθνικό και πολλές φορές και στο περιφερειακό και τοπικό. Κυρία Πονσελέ. Θα ήθελα απλώ να προσθέσω ένα σχόλιο για την κυρία Σιόντροβα. Το Erasmus Plus όντως είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ενθαρρύνει τη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό μας έχει επιτρέψει να δημιουργήσουμε για παράδειγμα, μια σχέση, μια εταιρική σχέση η οποία δεν θα υπήρχε χωρίς το Erasmus Plus και επίσης ακολουθούμε μια λογική πολιτισμού. Ξέρετε τι κάναμε το ε, μουσική για τους Ρωμά έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά στερεότυπα που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά σε όλη την Ευρώπη είναι μια ευρωπαϊκή διασυνοριακή μειονότητα με πολύ πλούσια παράδοση και μέσω αυτού δημιουργήσαμε ε, ένα ανθολόγιο, ένα ρεπερτουάρ για τους ε, δασκάλους για να μπορούν να διδαχθούν από αυτή ε, την κουλτούρα και να το χρησιμοποιήσουν και για άλλες. Δηλαδή τι μας έχει μάθει κάθε διαφορετική κουλτούρα, ποια είναι τα εργαλεία που είναι προσιτά για τους δασκάλους, για να αποκαλύψουν ε, την πλούτο μιας ε, ε, παράδοσης που θα μπορούσε να είναι η βερβερίνικη, η αρμένικη, συγκεκριμένη περίπτωση είναι η τσιγκάνικη των Ρωμά, μέσω κάποιων απλών ε, μέσων όπως τα μουσικά όργανα, για παράδειγμα, τα απλά, τα οποία χρησιμοποιούν παιδιά και τα οποία έχουν εμπνευστεί από την τσιγκάνικη μουσική. Τραγούδια, τραγούδια που τραγούδησαν μαζί γιατί ο τρόπος ε, που ε, τραγουδάνε οι Ρωμά ε, χρησιμοποιήθηκε για να εξοικειωθούν οι δάσκαλοι με τη γλώσσα αυτή, δεν τη μιλάνε πολύ αυτή τη γλώσσα. είναι όμως μια μεγάλη παράδοση, προέρχονται από την Ινδία, έχουμε τις παραδόσεις της Σαν Τη ε, της που βρίσκουμε στους Ρωμά στην Ισπανία. Άρα λοιπόν είναι κάτι που μπορούμε να μοιραστούμε όχι μόνο με τα παιδιά αλλά και με τους δασκάλους. Πιστεύω λοιπόν πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε με μια συνεχή εκπαίδευση των δασκάλων έτσι ώστε να ανακαλύπτουν τον πλούτο μιας παράδοσης που έρχεται να μας συναντήσει μέσω τέτοιου είδου project. Γι' αυτό χάρη στο Erasmus Plus που μπορέσαμε να το ε, στήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπεζότση. Euh, να τονίσω και να υπογραμμίσω και να δώσω έμφαση στο πόσο σημαντική ήταν η συζήτηση σήμερα το απόγευμα. Πρέπει οι διδάσκοντες να εμπνευστούν από την ιδέα ότι οι ίδιοι μπορούν να καλλιεργήσουν τη δημιουργία κοινωνικών δεσμών. Το σχολείο έχει επικεντρωθεί πολύ στην μάθηση και την επιτυχία στην μάθηση. Όμως υπάρχει το πολιτιστικό κεφάλαιο των μαθητών που περνάνε από τις αίθουσες διδασκαλίας. Πρέπει λοιπόν το σχολείο να δώσει μεγαλύτερη προσοχή και στο κοινωνικό κεφάλαιο που ε, μπορεί να καλλιεργείται στο εσωτερικό του και να επιτρέψει ανάπτυξη και εκτός σχολείου. Αυτό το σχολείο ακόμη δεν το καταφέρνει. Πρέπει να ανοιχθεί στην υπόλοιπη κοινωνία και να φανεί και να λειτουργήσει ως ένα αποστακτήριο του, της πεμπτουσίας της γνώσης που θα ε, γόνιμοποιήσει το έδαφος εκτός σχολείου. Το ίδιο και οι οικογένειες, οι γονείς και ένας κοινωνικός ιστός που διαρκώς αναδιαμορφώνεται. Εδώ λοιπόν ο κοινωνικός ιστός είναι η βάση της κοινωνικής ένταξης, είναι η βάση της παιδείας. Ιδάλλως δεν μπορεί να υπάρξει ένταξη. Μπορούμε να βρούμε όλα τα υπέροχα μοντέλα ένταξης που θέλουμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά πραγματική ένταξη γίνεται βάση της πράξης. Και δεν μιλώ μόνο για καλές διδακτικές πρακτικές, αλλά πρακτικές κοινωνικές, κοινωνικές συμπεριφορές. Δηλαδή το σχετίζεστε με κάποιον, το μοιράζεστε και συμμερίζεστε εμπειρίες, η αφοσίωση προσοχής, το στρέψιμο της προσοχής και κάτι που με ανησυχεί πολύ ως κίνδυνος που όλοι μπορεί να αντιμετωπίσουμε είναι η αποδυνάμωση, η αποδυνάμωση και η ένδυα του κοινωνικού ιστού, υποβάθμιση του κοινωνικού ιστού της Ευρώπης ολόκληρης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, ήταν πολύ γόνιμη η συζήτηση με πολλές αξιόλογες πληροφορίες και είναι σαφές ότι γνωρίζουμε όλοι ότι χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις αυτής της χωρίς προηγούμενο κρίσης προσφύγων στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε πολλές πολιτικές και όλες τις πολιτικές και εργαλεία στη διάθεσή μας και από πλευράς των θεσμικών οργάνων για τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές είναι επίσης σαφές ότι χρειαζόμαστε όλους τους εμπλεκόμενους κράτη-μέλη οπωσδήποτε, διότι δεν έχουμε εμείς τις αποκλειστικές αρμοδιότητες, έχουν τα κράτη-μέλη πολλές αρμοδιότητες στον τομέα του πολιτισμού, παιδείας και εκπαίδευσης. Θέλουμε να συνδυάσουμε και να μπορέσουμε να δράσουμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο βέβαια, αλλά χρειαζόμαστε και τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς και φορείς και χρειαζόμαστε και την κοινωνία των πολιτών, τις κοινωνίες επιτόπου στις διάφορες χώρες. Θα ήθελα να ανακεφαλαιώσω κάποια από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα από την απόψινή αυτή συνάντηση Πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να οικοδομήσουμε στο να εντάσσονται οι άνθρωποι και να ανήκουν σε ένα κοινωνικό περίγυρο και να μπορέσουν να προχωρήσουν έτσι. Το να ανήκει κανείς είναι θέμα κοινωνικής αρμοδιότητας και των δικών του επιδόσεων και πρέπει σε αυτό να οικοδομήσουμε και πρέπει έτσι να καταστήσουμε σαφές ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν και εκείνα περισσότερα ήταν πολύ ενδιαφέρον ε, βλέποντας ε, με τους καθηγητές και δασκάλους πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε να αντιμετωπίσουν καλύτερα όλα τα θέματα του πολιτισμικού διαλόγου και να προσφερθούν στα παιδιά δυνατότητες να μαθαίνουν αυτά τα πράγματα στα σχολεία μας. Χρειαζόμαστε αυτά τα μέσα και να υπάρξουν πρόσθετα κονδύλια. Χωρίς πρόσθετα κονδύλια δεν μπορούμε να επιτελέσουμε αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια που καταβάλλετε. Είναι σαφές ε, το τι πρέπει να γίνει σημαίνει και είναι απόλυτα κατανοητό και σαφές ότι χωρίς πρόσθετα κονδύλια δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό να ακούσουμε το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει πραγματογνωμοσύνη, ιδιαίτερα όσον αφορά την διαπολιτισμική εργασία σε σχέση με τους νέους. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ρατσισμό που ε, ε, υπάρχει και να δράσουμε ώστε τα θεσμικά όργανα και τα προγράμματα σε σχέση με τη δουλειά για τους νέους να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν με τρόπο ώστε να είναι αποτελεσματικά να έχουν τα μέσα στη διάθεσή τους δηλαδή η ένταξη η ένταξη ως κοινωνική δράση είναι κέρια σημασία επίσης διότι όλοι έχουμε καθήκοντα και ρόλο να αναλάβουμε ώστε η ένταξη είναι ένα κοινό έργο και εγχείρημα κοινή πρόκληση που πρέπει από όλους όλα τα κοινωνικά επίπεδα να αντιμετωπιστεί και τέλος αλλά εξίσου σημαντικό είναι να ε, συνειδητοποιήσουμε ότι οι τέχνες και τα οικαστικά βοηθούν, μπορούν να βοηθήσουν τους νέους, αλλά όχι μόνο τους νέους, να βρουν τη φωνή να εκφραστούν σωστά και να μπορέσουν να έχουν επαφή και να συνδεθούν με τις κοινωνίες προέλευσης τους αλλά και τις κοινωνίες υποδοχής. Αυτό που ξεκινήσαμε να κάνουμε με τα προγράμματα είναι αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε στη δράση μας ώστε να στεφθεί με επιτυχία αυτό το εγχείρημα. Για όλους αυτούς τους λόγους σας ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Ευχαριστώ τα μέλη του ακροατηρίου. Καλό σας βράδυ. Γεια σας και ευχαριστώ.